Η κυρία, Αϊάλα έχει καθυστερήσει έχει καθυστερήσει ένα ηφαίστειο στην Γουατεμάλα και ένας, ε, μια τροπική καταιγίδα στο Ελσαβαδόρ. Διαφορετικά θα βρισκόταν εδώ πέρα μαζί μας. Η δική μου λοιπόν η έκθεση που κανονικά είναι τελευταία στη μερίσια διάταξη θα είναι το πρώτο σημείο για το οποίο θα μιλήσουμε. Αυτά λοιπόν σας τα λέω προκειμένου να καταφέρουμε να εγκρίνουμε και την ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχει καμία παρατήρηση βλέπω. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έγκριση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης. Εγκρίνονται τα πρακτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τρίτο σημείο ανακοίνωση της νέας θέσης Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση στην Ολομέλεια της 18ης ε, Μαΐου στο Στρασβούργο σε πρώτη ανάγνωση η θέση του Συμβουλίου για την έγκριση της οδηγίας ε, για το πλαίσιο της εφαρμογής ευφυών συστημάτων μεταφορών στα πλαίσια των οδικών μεταφορών και για τη διεπαφή με άλλα μέσα μεταφοράς. Ανακοινώθηκε λοιπόν από το Συμβούλιο και υποβιβάστηκε στην Επιτροπή μας. Υποβλήθηκε, με συγχωρείτε. Λοιπόν, μετά τις ανακοινώσεις που γίνανε στην Ολομέλεια μου ζητήθηκε να σας ενημερώσω για τη θέση αυτή του Συμβουλίου. Κατ' επίσημο λοιπόν τρόπο πρέπει να το κάνω αυτό εδώ στην Επιτροπή μας. Θα θυμάστε ότι στην πρώτη ανάγνωση που εγκρίναμε στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου, ζητήθηκε από, το, από την συγκητή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για να επιτευχθεί συμφωνία στην δεύτερη ανάγνωση. Με την Σουηδική και την Ισπανική Προεδρία καταλήξαμε σε μία συμφωνία το Δεκέμβριο του 2009 και στις 10 Μαρτίου του 2010 στη συνέχεια και οι σχετικές πληροφορίες σας έδωσα σε επιστολή μου της 11ης Μαρτίου του 2010. Ενημέρωσα λοιπόν τα μέλη της ε, Επιτροπής για τις ε, συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Αν όχι, ας περάσουμε στο επόμενο σημείο της μερισσίας διάταξης. Στατιστικά δεδομένα μεταφορά αγαθών στατιστικά δεδομένα επιστροφής, μεταφορά αγαθών και επιβάτες στις θαλάσσιες μεταφορές. Στόχος της πρότασης αυτής είναι να τροποποιηθεί η οδηγία του 2009-42 προκειμένου η συλλογή δεδομένων να να γίνεται υποχρεωτικά η συλλογή δεδομένων ανατύπω προϊόντων και αυτό για τις θαλάσσιες μεταφορές. Η συλλογή αυτών δεδομένων γίνεται σε θελούσια βάση από 18 μόνο κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι πέντε κράτη-μέλη δεν έχουν θαλάσσιες ακτές και επομένως δεν υποβάλλουν δεδομένα στα πλαίσια της οδηγίας αυτής. Ως επιτοπλίστων η συλλογή των δεδομένων αυτών δεν πρόκειται να επιφέρει επιπλέον άχθο στα κράτη-μέλη και έτσι λοιπόν τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να συλλέγουν και να καταρτίζουν τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιώντας υφιστάμενους πόρους. Για παράδειγμα, τα έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούν οι λιμενικές αρχές ήδη. εισάγοντα όμως την υποχρέωση αυτή για τα στατιστικά δεδομένα θαλασσίων μεταφορών, όπως και για τα υπόλοιπα μέσα μεταφορών, δημιουργείται η υποχρέωση συλλογής δεδομένων προκειμένου να έχουμε μια απόλυτη συγκρισιμότητα ανάμεσα στα διάφορα μέσα μεταφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, η διαθεσιμότητα ομογενών και πλήρων στατιστικών δεδομένων ανατύπω αγαθού για όλα τα μέσα μεταφορών θα δώσει ένα εύχριστο γενικό πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να υποστηρίξουμε και να παρακολουθήσουμε, να επιτηρήσουμε καλύτερα την διατροπικότητα στα πλαίσια των ε, ευρωπαϊκών μεταφορών. Ως εισηγητής είμαι υπέρ της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν έχω να προτείνω καμία τροπολογία όσον αφορά την ουσία της πρότασης αυτής. Ωστόσο, η τροποποιημένη αυτή οδηγία παρέχει και κάποιες ε, αλλαγές όσον αφορά διαδικασία. Επομένως, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι ε, θα μπορούσαν να προσαρμοστούν οι νέες αυτές διατάξεις στο πλαίσιο των ε, κατεξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων που προβλέπει πλέον η συνθήκη της Λισαβόνας. Έχοντας λοιπόν αυτό κατά νου και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτίθεται να υποβάλει μια γενική πρόταση, μια οριζόντια πρόταση όσον αφορά τις κατεξοδότηση πράξης, προτείνω εγώ μια σειρά τροπολογιών για τις ε, κατεξοδότηση αυτές πράξεις, τις Delegated Acts. Ολοκληρώνω λοιπόν την παρουσίασή μου στο σημείο αυτό. Το λόγο μπορεί να πάρουν οι ο δισηγητές, ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ Κοιτάξτε, όσον αφορά statistical returns, carriage of goods and passengers, πράγματι έχετε δίκιο για πρώτη φορά να μπορούμε να πούμε ότι έχουν κατατεθεί τροπολογίες ε, και επιθυμούμε να ορίσουμε επακριβώς αυτό που αποκαλούμε delegated acts. Ως εκ τούτου κύριε Σίμψον, εμείς ως ΕΛΚ συμφωνούμε με αυτά τα οποία εσείς είπατε. και σας ευχαριστούμε για όλα αυτά τα τόσο σημαντικά που μας ε, παρουσιάσατε. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα αντικαταστήσω τον ε, συνάδελφό μου που δεν μπορεί να παρήσταστε και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε κύριε Σίμψον. Συγγνώμη που έπρεπε να παραγγείλω τον καφέ. Λοιπόν, συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που είπατε εσείς όπως και με την ε, πρόταση της ε, Κομισιόν και με τις απόψεις σας κατά την άποψη των φιλελευθέρων. Πρόκειται για θαυμάσιο έργο και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Η κυρία Κοιτάξτε, εγώ έχω να κάνω μία ερώτηση όσον αφορά στις ε, υποχρεώσεις ε, που έχουν ε, περιοχές που μπορούν να ερμηνευτούν ως ενδοχώρα. Δηλαδή, ερωτώ, ε, πού θα συγκεντρώνονται τα δεδομένα, προέρχονται από τις ε, εμπορικές συνταλλαγές, δηλαδή κάθε εταιρεία η οποία ε, αποστέλει ένα εμπόρευμα μέσω θαλάσσης υποχρεούται να το καταγράψει κάπου ή μήπω είναι δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται στα λιμάνια για να έχουμε μια σαφή εικόνα. Διότι εγώ διαπιστώνω ότι δυστυχώς πολλές φορές ε, δρομολογούνται περιττές διαδικασίες επί παραλήψη ε, παραδείγματος χάνει στην περίπτωση της Αυστρίας ε, υπήρξε μια ολόκληρη διαδικασία για δεξαμενόπλια διπλού, με διπλά τυχώματα. Άρα δηλαδή Νομίζω ότι εάν μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε με άλλο τρόπο τα δεδομένα, θα μπορούσαμε να αφήσουμε αυτή την περίπτωση της ενδοχώρας. Και ε, με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε λιγάκι σε επίπεδο ε, γραφειοκρατίας. Ευχαριστούμε κύριε Λίχτεμπεργκερ. Είπα και εγώ ότι πέντε κράτη-μέλη στερούνται ακτών. και πολλές τελωνιακές πληροφορίες χρειάζονται, αλλά ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να δώσει μια πιο ιδιεξοδική απάντηση, αν επιθυμεί. Δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο, οπότε υπάρχει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα αυτό. No. We have nobody from the Commission to answer your question, so your best answer is going to... Οπότε, δυστυχώς, εγώ θα απαντήσω, Εύα. Άλλη πιο έγκυρη απάντηση δεν θα έχετε για τα στατιστικά. Τις στατιστικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα τελωνία και κάποιες οργανισμούς που είναι αρμόδιοι με τον έλεγχο των εφαρμογ... της εφαρμογής, τότε ας μας στείλει γραπτό στην απάντηση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής γιατί θα μας διαφωτίσει και στην όλη συζήτηση κατά της γραφειοκρατίας. Καλώς, θα το ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια γραπτή απάντηση. Καλώς. Πολύ γρήγορα διεκπεράσαμε αυτό το θέμα και μπορούμε να πάμε στα δικαιώματα των επιβατών, λεωφορείων και πούλμαν. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες, αλλά να σας υπενθυμίσω την 3η Ιουνίου που λύγει η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. 22 Ιουνίου θα, πάει στην, θα ψηφιστεί στην Επιτροπή μας και κατά πάσα πιθανότητα στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Κατά προτίμηση στην πρώτη, θα δούμε. Ίσως δεν προλάβουμε στην πρώτη. Επόμενη έκθεση του κυρίου Κάντσαν. Δικαιώματα των επιβατών, λεωφορείων και πούλμαν. Κύριε Καντσάν, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις εισηγητές, ε, κυρίως ε, τις τρεις συναδέλφου, Τσερκιάνη, ε, Μάισνερ και Λίχνμπεργκερ οι οποίε ε, παρακολούθησαν ε, πολύ πιο πολύ εκ του περισσότερο και από μένα όλη αυτή τη δουλειά και με βοήθησαν επί της ουσίας πραγματικά με συνέδραμαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και Επίσης ε, θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για θέματα μεταφορών. Κοιτάξτε, βλέποντας αυτή την έκθεση νομίζω ότι είναι σημαντικό να επενθυμίσουμε ότι η θέση του Συμβουλίου στην πρώτη ανάγνωση ε, είναι απαράδεκτη, διότι υπάρχουν πολύ σημαντικοί περιορισμοί όσον αφορά τους ε, προβλεπόμενους ε, στόχους ε, και τις εξαιρέσει για εκείνου που παραμένουν μέσα στους στόχους. Μιλάμε για αυτά τα 15 χρόνια απαράδεκτη και διότι υπάρχουν εξαιρέσει όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιπε διατάξεις και αυτές αποδυναμώνονται αδικαιολόγητα. Εάν λοιπόν εγκριθεί η θέση του Συμβουλίου, τότε δεν θα αλλάξει τίποτα σε σχέση με αυτό που ισχύει τώρα δηλαδή αυτό είναι απαράδεκτο όσον αφορά την προστασία των επιβατών. Η δική μου λοιπόν η σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση βασίζεται στην πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και θέλω να σα το επενθυμίσω εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία κατά τη διάρκεια τη ολομέλεια, ακριβώς όπως αναφέρεται στην επεξηγηματική έκθεση του σχεδίου σύσταση. Εξηγήθηκε επίση ε, το πλαίσιο εφαρμογή ε, ο χρόνο εφαρμογή, ε, η

οι ευθύνε προφανώς ε, όπως επίσης ε, και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και με περιορισμένη κινητικότητα. Εγώ ε, θέλω να θεωρήσω ότι να πω ότι τα δικαιώματα των επιβατών πρέπει να γίνουν αποδεκτά και αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό από όσους προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες λεωφορείων και πούλμαν. Η δική μου λοιπόν η πρόθεση είναι να υπάρχει κάποια εξισορρόπηση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές θέσεις αντίθετες θέσεις. Και όσον αφορά τι διαπραγματεύσει, θέλω να πω ότι πραγματικά ήταν πολύ καλή αυτή η εμπειρία συνεργασία που κάναμε. Εγώ τη δική μου τη θέση την έχω συντονίσει με τη θέση των ε, ε, εισηγητών, ε, των σκιωδών εισηγητών και είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία, κυρίω την τελευταία μας συνάντηση όπου καταλήξαμε σε μια κοινή θέση για τα σημαντικά θέματα. Του τελευταίου μήνε είχαμε διάφορες τριγωνικέ συζητήσει με την Ισπανική Προεδρία με την οποία είχαμε μια πολύ επικοδομητική σχέση και βρήκαμε, καταλήξαμε σε ε, ρεαλιστικά, ε, ρεαλιστικές προτάσεις. Και αυτό βέβαια γιατί συνέβαλε και η Επιτροπή σε όλο αυτό. Συμφώνησα λοιπόν με τους σκιώδη ηγητές μία σειρά από προτάσεις συμβαστικές. Συμφώνησα και με το Συμβούλιο για τα πιο σημαντικά θέματα που είναι κυρίως όσον αφορά το πλαίσιο των ε, ευθυνών και των αρμοδιοτήτων. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ισπανική Προεδρία πρέπει να επιδείξει την απαραίτητη ευελιξία έτσι ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αυτά που ακούμε τώρα τελευταία από το Συμβούλιο δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Γιατί αντί το Συμβούλιο να μετακινηθεί προ εμά, προ το Κοινοβούλιο, έκαναν και μισό βήμα προ τα πίσω. Είναι λοιπόν το Συμβούλιο να προχωρήσει σήμερα το βράδυ, κατά τη διάρκεια τη τριμερού αυτή συζήτηση που έχουμε προβλέψει και ε, με στόχο να μπορέσουμε τελικά να καταλήξουμε σε ένα αίσιο τέλος. Βεβαίω, ε, έχοντα υπόψη αυτά που είναι γνωστά, είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή μα να δώσει ένα σαφέ δείγμα υποστηρίξη και να εγκρίνει, να υιοθετήσει την έκθεση με σαφή πλειοψηφία, έτσι ώστε να δοθεί σε μένα και στου και ηγητές μια σαφή εντολή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τι διαπραγματεύσει. Και τέλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω και για τι πολύ επικοδομητικέ τροπολογίες που έλαβα εκ μέρου ορισμένων συναδέλφων. ορισμένε ε, εξ αυτών συμπληρώνουν τη δικαιοσύνη δική μου τη θέση και καθίσταται η θέση μας περισσότερο σαφής. Άλλες πάλι αναγκάστηκα να τις απορρίψω, κυρίως εκείνες ε, ε, που ε, δεν με βοηθούν στο να διατηρήσω τη δική μου την τελευταία θέση που κατέθεσα στο Συμβούλιο. Αυτό το βλέπετε στην προφορική τροπολογία που καταθέσει την υπαριθμών 11. Επίσης ε, θεωρώ ότι όσον αφορά τη χρονική στιγμή είναι κατάλληλη αυτή η χρονική στιγμή γιατί αν καθυστερήσουμε κατά την άποψή μου υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστούν επικίνδυνες συμπεριφορές εκ μέρους των ε, ε, οδηγών. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε τη συζήτηση και αύριο την ψηφοφορία που θέλω να πιστεύω ότι θα οδηγήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε κύριε Κάντσαν. Από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ε, κυρία Σαρετσιάνη ζήτησε το λόγο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστώ τον κύριο Κανσιάν για την πολύ καλή δουλειά που παρουσίασε, που ήταν και πραγματικά πολύ χρήσιμη. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να υπογραμμίσω τα σημαντικότερα θέματα για τα οποία από με του ε, συναδέλφου μου αγωνιστήκαμε για τα δικαιώματα των επιβατών, λεωφορείων και πούλμαν. Ε, στο θέμα που ενδιαφερθήκαμε για συμβασμό είναι κυρίω το πεδίο εφαρμογή. Η πρόταση στην πρώτη ανάγνωση εγκρίθηκε πέρυσι και πρόκειται για μια πολύ σωστή εφαρμογή για όλα τα μέσα μεταφορά ε, τα κράτη-μέλη λοιπόν έχουν την ε, δυνατότητα να εξαιρούν περιφερειακές μεταφορές όταν αυτές δεν καλύπτονται από ε, την δέουσα προστασία. Εγώ λοιπόν συμφωνώ ότι πράγματι πρέπει να είναι δυνατόν να εξαιρούνται μόνο οι περιφερειακές μεταφορές όταν βέβαια υπάρχει κάποιο δίκτυο αστικό. Όσον αφορά το θέμα των αρμοδιοτήτων, κυρίως το θέμα των προκαταβολών. Εκεί θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο συνετοί με στόχο να μην υπάρχει κίνδυνος απατών. Γιατί όσον αφορά τις προκαταβολές αυτές θα πρέπει να μπορούν να επιστραφούν πάρα αυτά για να μην υπάρχει κίνδυνος απάτης και ε, θα έπρεπε να αποκλειστεί μάλιστα αυτό ο κίνδυνο στα διάφορα κρατημέλη. Υπάρχουν και διαφορετικές ε, ασφάλειες ε, όσον αφορά την αστική ευθύνη. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι πρέπει να γίνεται αναφορά στην εθνική νομοθεσία της χώρας όπου λαμβάνει η χώρα ένα συμβάν. Το άρθρο 21 προβλέπει την υποστήριξη όταν υπάρχει καθυστέρηση πάνω από δύο ώρε. Στην περίπτωση αυτή καλύτερα να λέμε η καθυστέρηση καθυστέρηση μια ώρα και όχι δύο ώρων για τα δικαιώματα των επιβατών. Και έτσι οι επιβάτε να έχουν τα ίδια δικαιώματα όπω και με άλλα μέσα μεταφορά, όπω με το τρένο. Ε, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιστροφή των χρημάτων του 50% του στηρίου σε περίπτωση ε, καθυστέρηση πάνω από δύο ώρε, Εφόσον βέβαια η ε, καθυστέρηση οφείλεται στο πούλμαν. Όσον αφορά το άρθρο 24, στην παράγραφο 1 στα δικαιώματα των επιβατών, εκεί είναι σωστό να λέμε ότι οι επιβάτε πρέπει να ενημέρονται για την ε, διαλειτουργικότητα και νομίζω με τον τρόπο αυτό θα ε, διασφαλιστεί ε, και η εύρυθμη λειτουργία όλων των μέσων μεταφοράς. Όσον αφορά τώρα τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα πρέπει να υπάρχει η μέγιστη προστασία 24 ώρες να λέμε και όχι 48 ώρες έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρεται η υποστήριξη. Όσον αφορά τώρα την ε, κινητικότητα σε περίπτωση απώλειας ζημιάς. Ε, εκεί θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα δικαιώματα των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Μην υπάρχει κανένας φραγμός να διευκολύνονται τα άτομα αυτά. Ε, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Thank θα ήθελα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ε, τον τρόπο με τον οποίο ε, συζητήσατε μέχρι τώρα στην ε, τριμερή συζήτηση. Δύσκολη συζήτηση. Πολύ καλό αυτό που είπατε διότι το Συμβούλιο προφανώς εμένει στις θέσεις του. Και ε, πράγματι επιτύχαμε πολλούς συμβασμούς και προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε μια κοινή γραμμή. Ε, ελπίζαμε όλοι ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν κάτι τέτοιο και ελπίζουμε στο μέλλον να συνεχιστεί η διαδικασία. Ελέγχθησαν πολλά. Κατά την πρώτη ανάγνωση υπήρξε αμέριστη υποστήριξη αυτών που παρουσιάστηκαν και εμείς ε, προσανατολιστήκαμε σε αυτή την πρώτη ανάγνωση. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εκ μέρους των φιλελευθέρων υποστηρίζω ακριβώς αυτά που ο κύριος Κάντσα θέλουμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των επιβατών. Παράλληλα βέβαια να αναζητήσουμε το τι είναι εφικτό, τι μπορούμε να περιμένουμε από επιχειρήσεις που προσφέρουν πούλμαν, γιατί μην ξεχνάτε ότι εδώ πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρέπει να μπορούν να λειτουργούν και στο μέλλον. Αυτό λοιπόν ήταν μια σκέψη, ένα οδηγό νήμα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Τώρα, όσον αφορά τις αρμοδιότητες, εξακολουθεί να μην έχει αποφασιστεί ποιο θα είναι αρμόδιο. Το Συμβούλιο λέει ναι, να εξαιρεθούν οι περιφερειακές ε, μεταφορές. Ναι, και εμείς συμφωνούμε μόνο όμως εφόσον υπάρχει διασύνδεση με αστικές ε, μεταφορές, όχι σε άλλη περίπτωση. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν συμφωνήσαμε επ' αυτού. Όσον αφορά τώρα την ενημέρωση, η συνάδελφη κυρία Αρκιάνη τοποθετήθηκε επ' αυτού, αλλά πράγματι είναι απαραίτητο ε, να υπάρχει μια διαφάνεια στις πληροφορίες και για άτομα με αναπηρία. Αυτό να το προσέξουμε και να μην ενδώσουμε σε αυτό. Όσον αφορά την αποζημίωση, ε, πράγματι τι ε, μένεται η μάχη με το Συμβούλιο και θα δούμε τελικά πού θα τοποθετηθούμε εμείς. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι όσον αφορά τις ε, τροπολογίες εμείς θα θέλαμε ε, ψηφοφορία σε τμήματα στην τροπολογία υπαριθμών 40 παρακαλώ αν γίνεται. Να ψηφίσουμε σε δύο τμήματα την τροπολογία αυτή. Αυτά εκ μέρους πολιτικής μου ομάδας. Σας ευχαριστώ κύριε Κάντσα για την εργασία σας και βέβαια θα συνεχίσουμε με αυτό το αγώνα που δίνουμε. Η κυρία Λίχτιμπεργκα. Ε, ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Κάντσα για την ε, δέσμευση και στράτευση που επέδειξε για το θέμα αυτό. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είμαι εξοργισμένη με τη στάση του Συμβουλίου. Κυρίως όσον αφορά στα θέματα, στα δικαιώματα επιβατών με αναπηρία. Το να είναι τόσο σκληρό το Συμβούλιο, ε, για μένα αυτό είναι ακατανόητο. Γιατί όπως πολύ σωστά ελέγχθη, για αυτούς τους ανθρώπους ε, δεν θα υπάρξει καμία θετική αλλαγή αν τελικά η συμφωνία κλείσει όπως τη θέλει το Συμβούλιο. Και για μένα αυτό είναι απαράδεκτο γιατί υπάρχει η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και αυτό βέβαια ισχύει και για τον ε, τομέα των μεταφορών και πρέπει να ισχύει εκεί, πόσο μάλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι το να γίνεται αυτή η διαφοροποίηση των ε, περιφερειακών και των αστικών μεταφορών. Όπως το είπα και την τελευταία φορά, οι ε, περιφερειακές αυτές ε, μπορεί να είναι και μακράς διάρκειας. Ε, μπορούν να φορούν μεγάλες αποστάσεις μπορούν να είναι πολύ σημαντικές σε κάποια κρατημέλη όπου οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι απαράδεκτες ή δεν υπάρχουν άλλα μέσα μεταφοράς. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να εξευρεθεί ε, ένα συμβαστικός τύπος ε, που να αφορά στα δικαιώματα των αναπήρων στις υπεραστικές μεταφορές. Να ε, αναγνωρίζονται τα δικαιώματά τους τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν ε, δικαιώματα ατόμων με αναπηρία σε κάποιες εθνικές νομοθεσίες. Αυτό που επίσης έχει σημασία είναι οι πληροφορίες ε, για τα εισιτήρια, για τα ωράρια, να είναι προσπελάσιμες. Αυτό είναι καθοριστική σημασία. Πρέπει λοιπόν να κατορθώσουμε τα δικαιώματα των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα να τα ενισχύσουμε όπως επίσης και να ενισχύσουμε το δικαίωμα στην ενημέρωση για όλες τις μορφές αναπηρίας. Γιατί όλα αυτά με τη σημερινή τεχνολογία είναι εύκολο να προσφερθούν και δεν είναι και δαπανηρά, αλλά ακόμα και αν ήταν δαπανηρά πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Επειδή λοιπόν παρουσιάζεται γύρανση στον πληθυσμό μας, θα έχουμε όλο και περισσότερο τέτοιους πολίτες. Και γι' αυτό παρακαλώ εσείς στο Συμβουλίο να το λάβετε αυτό υπόψη σας. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την απαράδεκτη αντίδραση απέντησε θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, Mr. E Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπράντμπορν για τους μεταρρυθμιστές και συντηρητικούς. Στην πρώτη συζήτηση για το θέμα αυτό είπαμε ότι η προσπάθεια αξιέπαινει και το σχέδιο, αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και μετά την ανάγνωση γνωμοδότηση επιβεβαιώθηκε αυτή η άποψή μου. Εδώ δεν έχουμε ίση μεταχείριση. Όταν μιλούσαμε για τα δικαιώματα των αεροπορικών μεταφορών των σιδηροδρομικών, μιλούσαμε για επιβάτες που είχαν να αντιμετωπίσουν μεγάλες οργανώσεις και παρόχους υπηρεσιών, αλλά στα λεωφορεία και τα πούλμον, το 85% των εταιριών, των επιχειρήσεων που εξασφαλίζουν αυτές τις μεταφορές είναι μικρομεσαίες. Δεν είναι οι κολοσσιαίες επιχειρήσεις όπως σε αερομεταφορές, οπότε και η αντίδραση που θα πρέπει να δώσουμε και η απάντησή μας στην πρώτη Συμβουλή και της Επιτροπής θα πρέπει να είναι ανάλογη με αυτές τις διαστάσεις. Με τις τροπολογίες μου προσπάθησα να προσαρμόσω και να προσγειώσω στην πραγματικότητα τις ε, προτάσεις αυτές και τι είναι εφικτό στις συμφωνίες μας με το Συμβούλιο. Και από αυτή την άποψη θα πρέπει πολύ προσεκτικά να εξετάσουμε τις τροπολογίες που ουσιαστικά ζητούν παρόμοια ρύθμιση με αυτή που ισχύει για τις ε, μεγάλες εταιρείες και μεγαλύτερες οργανώσεις. Θα αναφερθώ σε ορισμένα τα θέματα αυτά. Καταρχήν, το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Εδώ εξετάζουμε το είδος των υπηρεσιών που θα πρέπει να καλύπτονται από την πρόταση αυτή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει γενικό τεκμήριο για αυτοεξαίρεση των κρατών μελών από την πρόταση αυτή όταν έχουν το δικό τους τρόπο εφαρμογής για τις περιφερειακές κυρίως συγκοινωνίες ή τις ε, συγκοινωνίες στις αγροτικές περιοχές, γιατί εκεί είναι που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξασφαλίζουν αυτές τις, μετε... τις υπηρεσίες. Και πολύ φοβούμαι ότι αν ε, ρυθμίσουμε με την παραμικρή λεπτομέρεια όλο αυτό το τομέα, θα εξαφανιστούν οι επιχειρήσεις αυτές από τις αγροτικές περιοχές. Δεύτερη μου παρατήρηση για την αποζημίωση και τις διάφορες διατάξεις της πρότασης για τις προκαταβολές και ούτω καθεξής. Και πάλι, επί της αρχής, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση εφόσον κάτι πάει στραβά ή εφόσον ακυρώνεται μία μεταφορά ή υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά δεν θα πρέπει να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, γιατί είναι ιδιάζουσα η κατάσταση στις μεταφορές με ολοφορία και πούλμαν. Εγώ διάβασα πολλές τροπολογίες και μερικές φορές προεξοφλούμε τη σωστή διαδικασία ε, ή τη σωστή δίκη, γιατί μιλούμε για προκαταβολές που αν ήταν σοβαρά τα τροχέα με λεωφορεία και πούλμαν, θα υπήρχε μια διαδικασία ε, νομική. Οπότε θα πρέπει να σεβαστούμε αυτή την ε, δικαστική οδό. Και εκεί, εδώ ισχύουν τα ένομα εθνικά συστήματα και οι εθνικές δικονομίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Θα ήθελα να επιθυμήσω στην Επιτροπή ότι και στο σιδηροδρομικό πακέτο εγώ ήμουν ε, ένθερμος υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ανθρώπων με μειωμένη κινητικότητα ή με ειδικέ ανάγκες για τις υπηρεσίες αυτές. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην ανάγκη ρεαλισμού και περιορισμού μας στο εφικτό. Τι μπορούν να προσφέρουν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι. Ορισμένες τέτοιες επιχειρήσεις θα πρέπει να προσφέρουν αυτές οι επιπλέον υπηρεσίες με χαμηλό κόστος ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αν το καταφέρουν αυτό με μικρό κόστος και όχι με θυσία την επιβίωσή του, συμφωνώ. Αλλά όχι να τις εξωθήσουμε σε χρεοκοπία μόνο και μόνο για να στενιστούν αυτές τις νέες διατάξεις, γιατί έτσι θα πληγούν όχι μόνο οι άνθρωποι με μειωμένη κινητικότητα γιατί θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες, αλλά και όλος ο υπόλοιπος κόσμος γιατί θα καταργηθούν αυτές οι υπηρεσίες, μια και θα πτωχεύσουν οι αντίστοιχε επιχειρήσεις. Μπράτμπορν. αλλά λάθος έκανα το όνομά γιατί έτσι, είναι, έτσι λέγεται ο κουνιάδος μου. Η κυρία Γιέγκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you very... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Κάντσαν καθώς επίσης και τους κοιόδης εισηγητές για την πολύ καλή δουλειά που έχουν κάνει στο θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να προστατευτούν περισσότερο οι επιβάτες και θεωρούμε ότι ε, ο σημερινός τριμερής διάλογος θα είναι μία ακόμα ευκαιρία για να βρούμε μια ισορροπημένη λύση και για να καταφέρουμε να καταλήξουμε συμφωνία. Θεωρούμε ότι και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σημαντικό δύο προτάσεις, όχι μόνο αυτές που έχουν να κάνουν με τα λεωφορεία και τα πούλμαν, αλλά και μια πρόταση που θα έχει να κάνει με τις θαλάσσιε και τις εσωτερικέ πρωτές μεταφορές θα πρέπει να εγκριθούν σύντομα και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να καλύψουμε το χάσμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην νομοθεσία και θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε όλου του επιβάτε σε όλο το φάσμα των μεταφορών συμπληρώνοντας έτσι τα όσα έχουν ήδη γίνει για το σιδηροδρομικό τομέα. Προσβλέπουμε λοιπόν σε ένα πολύ θετικό τριμερή διάλογο σήμερα το βράδυ και θα προσπαθήσουμε εμεί να διευκολύνουμε την έβρεση συμφωνίας. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Γέγκε. Κύριε Κάνσεν, έχετε το λόγο. Grazie, ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που ελέγχθησαν. Ο συνήθω είναι όλα πολύ, τα σχόλια ήταν επικοδομητικά και ελπίζω ότι τα περισσότερα από αυτά που ελέγχθησαν ελπίζω ότι σήμερα το βράδυ στη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου θα ληφθούν υπόψη. Τώρα, αυτά που ε, κατά την άποψή μου ε, πρέπει να εξεταστούν ενδελεχέστερα είναι κυρίως το θέμα της καθυστέρησης. Ο... Αναφέρθηκε ο συνάδελφος Τσαρακιάνη επί του θέματος αυτού. Κοιτάξτε, όσον αφορά την καθυστέρηση δεν ελέγχθη τίποτα. Εμείς ε, βέβαια εστιάζουμε την προσοχή μας στην αναχώρηση γιατί αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όσον αφορά όμως την άφηξη Εκεί πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο. Πολλές φορές οι οδηγοί ε, έχουν κάποιες ιδιαίτερες διαδικασίες που εφαρμόζουν για να μην καθυστερήσουν. Εκεί είναι λιγάκι αυτό που με απασχολεί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά που είπε η κυρία Τσαρακιάν τα λάβαμε υπόψη μας. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι. Όσον αφορά την ε, τα σχόλια της κυρίας Μάισνερ συζητήσαμε πολλές φορές ε, για την αποζημίωση και την επιστροφή των χρημάτων. Νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα και τις ε, τροπολογίες για το άρθρο 40 μπορούμε πράγματι να τις ψηφίσουμε σε δύο τμήματα, κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά τώρα την ε, παρέμβαση ε, κυρία Λίχτενμπεργκ από τους ε, Πράσινους νομίζω ότι έχει επιμείνει πάρα πολύ στο θέμα των δικαιωμάτων των ατόμων ε, με περιορισμένη κινητικότητα. Και εμείς συμφωνούμε απόλυτα από αυτού γιατί στην περίπτωση αυτή προφανώς είναι ο πρώτος μας στόχος άρα δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε βέβαια στο πλαίσιο των ορίων που υπάρχουν. Και το θέμα ε, της ενιαίας έκδοση και αυτό το θίξαμε για να είναι τα πράγματα λίγο πιο απλά. Και εκεί είναι τα χέρια μας λιγάκι δεμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά την του ε, αδέλφου Μπάντμπουρ, νομίζω ότι θα πρέπει να προβάλλουμε περισσότερο ορισμένα πράγματα. Εμείς προσπαθήσαμε να επιτύχουμε μία ισορροπία, το είπα και προηγουμένως, ανάμεσα σε αυτά που είναι τα δικαιώματα που αναφέρονται στην έκθεση, να τα ισορροπήσουμε αυτά με τα δικαιώματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί προφανώς δεν θέλουμε ούτε να γονατίσουμε τις επιχειρήσεις, ούτε να δημιουργήσουμε κανένα δικαιολόγητο πρόβλημα. Ούτε εγώ, ούτε και κανένας άλλος. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους πρόθεση. Βεβαίως αν μετακινηθούμε λιγάκι προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, τότε η ισορροπία θα διαταραχθεί γιατί ε, σε κάποιες περιπτώσεις το ένα δεν μπορεί κανείς ε, να το αγγίξει, το άλλο δεν προβλέπεται. Έχουμε τις αστικές μεταφορές, τις προαστιακές, ίσως ε, τις περιφερειακές. Μετά έχουμε κάνει διαχωρισμό ανάμεσα σε εσωτερικές, τακτικές, μη τακτικές διεθνείς μεταφορές. Τι έχουμε χωρίσει σε τέσσερις κατηγορίες τις μεταφορές, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να ρυθμίσουμε και τα θέματα του ωραρίου. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι σε αυτήν εδώ την περίπτωση το βάρος δεν πάει τόσο στα δικαιώματα των ε, πολιτών αλλά ε, περισσότερο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, Πάντως ε, εγώ θεωρώ ότι πράγματι πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο στα δικαιώματα των πολιτών γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή κλείνει προς την άλλη κατεύθυνση. Σήμερα το βράδυ έχουμε μια πολύ σημαντική τριμερή συζήτηση και έχω βάσιμες ελπίδες ότι στο πλαίσιο αυτού αυτής της συζήτησης θα μπορέσουμε να καταλήξουμε. Βεβαίω έχουμε και χρόνο μέχρι την ολομέλεια του Ιουλίου και μπορούμε ακόμα να εργαστούμε. Αλλά θα ήθελα έστω σήμερα, αύριο, να εκπέμψουμε ένα ηχηρό μήνυμα προ την Κομισιόν, προ αυτή την κατεύθυνση που σα εξέθεσα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάντσιαν. Να επαναλάβω τα όσα είπατε. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να πάμε στην Ολομέλεια τον Ιούλιο με την έκθεση αυτή. Το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη είναι η διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων. Η έκθεση της κυρίας Ντεβεράκ. Πιο νωρί από ό,τι προβλεπόταν η κυρία Ντεβεράκ αντιμετωπίζουμε το ζήτημα αυτό. Είστε έτοιμοι να μιλήσετε για την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τις τροπολογίες που υποβάλατε και σας ευχαριστώ που δεν υποβάλατε τόσες πολλές όσες είχαμε και στην έκθεση του κυρίου Μάθιου Γκρός που είχαμε φτάσει τις 400 περίπου τροπολογίες. Είμαι ως επιτοπλίστων υπέρ των τροπολογιών σας Αντί όμως να αφαιρθώ σε αυτές μία προς μία, θα ήθελα να αναφερθώ στις μεγάλες προτεραιότητες του κειμένου, καθώς επίσης και στις τροπολογίες τις οποίες απορρίπτω και θα τελογίσω βέβαια και την απόρριψή μου αυτή. Γενικά λοιπόν πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι για τις μεγάλες κατευθυντήρες γραμμές και τους βασικούς στόχους που θέλουμε να έχει ο νέος αυτός καονισμός. Όλοι επιθυμούμε έρευνες για τα ατυχήματα, αποτελεσματικές έρευνες που θα γίνονται από ικανές και αρμόδιες αρχές διερεύνησης που θα λειτουργούν αποτελεσματικά. Οι αρχές αυτές διερεύνησης θα μπορούν να βασίζονται στις ε, εθνικές αρμόδιες αρχές. Κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να καλύψουμε και τις, ε, την απόκληση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και να έχουμε 27 αρχές διερεύνησης οι οποίες είναι αποτελεσματικές και 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συγκεκριμένε αναφορέ αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει με τι αναφορέ να είμαστε σε θέση να μπορούμε να κάνουμε ανάλυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μπορούμε εκ των προτέρων να δούμε ποιε είναι αναδυόμενε τάσει και κατά αυτόν τον τρόπο να καταφέρουμε να αποφύγουμε και ορισμένα ατυχήματα. Τουλάχιστον αυτό είναι το ευκταίο για το μέλλον. Επίση, ελπίζω ότι μέσω του κανονισμού αυτού θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο ασφάλεια στι ε, αεροπορικέ μεταφορέ και είναι μια καταπληκτική ευκαιρία που δεν μπορούμε να τη στερήσουμε από τον Ευρωπαίο πολίτη. Καταλαβαίνω την τροπολογία 68 του ε, Προέδρου, την ε, υποστηρίζω, αλλά μόνο εφόσον μπορεί να συμπληρώσει τις δικές μου τροπολογίες για τις αναφορές για τα διάφορα συμβάντα. Συμφωνώ ότι θα πρέπει η οδηγία 43 του 2003 να μας επιτρέπει να κάνουμε τη σωστή ανάλυση, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε να κάνει νέα πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να τύχει διαπραγμάτευση η πρόταση αυτή, να υιοθετηθεί και να μεταφερθεί, για να λάβουμε εμεί δράση για την ανάλυση των δεδομένων που έχουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων ΕΚΕΡΣ. Χάνουμε πάρα πολλά χρόνια, χάνουμε πάρα πολύ χρόνο και συνδέουν διάφορα αεροπορικά ατυχήματα τα οποία αναφέρονται, ε, έχουν να κάνουν με διάφορε διαφορετικέ παραμέτρου. Διακόπτει ο Πρόεδρο. Κυρίε και κύριοι, υπάρχει πάρα πολύ στόρυβο μέσα στην αίθουσα. Πολλοί συζητούν μεταξύ του, πολλοί μετακινούνται μέσα στην αίθουσα. Αν θέλετε να μιλήσετε με κάποιον συναδελφό σα, κάντε το εκτό αιθού σα, παρακαλώ, έτσι ώστε η συγγήτρια και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να σε θέση να μιλήσουν και να παρακολουθήσουν τη συζήτηση τη έκθεση. Ε, αν θέλετε λοιπόν να μιλήσετε, κάντε το εκτό σα. Μπορείτε να συνεχίσετε, κυρία Ντεβέιρακ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είδατε επίση ότι είμαι βραχνιασμένη. Πρέπει λοιπόν να δράξουμε την ευθύνη αυτή που έχουμε με, την, με τον νέο αυτοκανονισμό και να ζητήσουμε τα δεδομένα που βρίσκονται στο κέντρο βάσης ΕΚΕΡΣ να αναλυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά τώρα την βοήθεια, την αρρωγή προς τα θύματα και προς τους οικείους τους, πάλι θεωρώ ότι οι ισχύουσες διατάξεις δεν αρκούν και μέσα από τον νέο κανονισμό μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο τα θύματα και τους οικείους τους. Όσον αφορά τώρα τον κατάλογο, αποκλίνει εδώ πέρα οι θέσει. Η κυρία Αλβάρη ε, θα θέλω ο κατάλογο αυτό μέσω τη τροπολογία 51 να είναι διαθέσιμο πριν την αναχώρηση. Η κυρία Τικάου με την τροπολογία 52 προτείνει ένα χρονικό διάστημα μισή ώρα. Εσεί κύριε Πρόεδρε ζητάτε δύο ώρε, 153 και 154 τροπολογίε. Εγώ προτιμώ να διατηρήσουμε την προθεσμία της μίας ώρας, μου φαίνεται λογική και άλλωστε έχει λειτουργήσει στην πράξη τόπου η διάταξη αυτή τώρα όσον αφορά την ε, συμμετοχή στις έρευνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΙΚΑΟ θα πρέπει όντως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Αεροπορίας να συμμετέχει στις έρευνες που γίνονται. Επομένως δεν μπορώ να υποστηρίξω τροπολογίες 114, 115 και 116. Οι δύο τελευταίες κυρία Πάρα πολλές τροπολογίες υποβλήθησαν και έχουν να κάνουν με τον ορισμό Έχουμε μία διεθνή νομοθεσία όσον αφορά τις ε, έρευνες για τα αεροπορικά ατυχήματα. Πρόκειται για το παράρτημα 13 που έχουμε στα πλαίσια του οργανισμού ΙΚΑΟ. Και ε, ακολουθούμε ουσιαστικά τον ορισμό αυτό, διαφορετικά θα προκληθεί μεγάλη σύγχυση. Σε περίπτωση λοιπόν ατυχήματος ακολουθούνται οι ορισμοί αυτοί και δεν θα έπρεπε νομίζω να αποκλίνουμε από το εφιστάμενο καθεστώς. Γι' αυτό το λόγο δεν υποστηρίζω τις ε, τροπολογίες αυτές προτείνουν άλλους ορισμούς πέρα από αυτούς προβλέποντας το παράρτημα 13 αναφέρουμε στις τροπολογίες 93-94 ε, 95 και 129, 72 και 99, 90, 92, 96 της κυριατικά, και τέλος 123. Αυτές είναι οι τροπολογίες τις οποίες δεν μπορώ να υποστηρίξω. Όσον αφορά τώρα τις έρευνες που γίνονται από τους αρμόδιους οργανισμούς αρχές διερεύνησης των κρατών μελών, καθώς επίσης και τις δικαστικές έρευνες που διεξάγονται από τα κράτη-μέλη, πιστεύουν το σημείο αυτό που δεν θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε πολύ εύκολα με το Συμβούλιο, γιατί εδώ πέρα έχουμε κάποιες τροπολογίες που ε, αντιτάσσονται στη θέση του Συμβουλίου και περιορίζουν ουσιαστικά την πρόσβαση της δικαιοσύνης στα δεδομένα τα οποία συλλέγονται στα πλαίσια των ερευνών ασφαλεία. Υποστηρίζω πολλέ από τις σχετικές τροπολογίες και πιστεύω ότι θα μας επιτρέψουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε ρυθμίσεις που θα μας επιτρέπουν με πολύ σαφή τρόπο να διαχωρίζουμε τα εμπιστευτικά δεδομένα και αυτά τα οποία μπορούν να πάνε στη δικαιοσύνη. Η τροπολογία 40 αναφέρεται στα στοιχεία αυτά. Επιπλέον σε κάθε κράτο μέλο θα πρέπει να έχουμε συμφωνίες ε, χρηστής συνεργασίας ανάμεσα στις αρχές διερεύνησης και τις δικαστικές αρχές. Έχω την τροπολογία επίσης 124 που συμπληρώνει την 126 και την 127 του Γέλκο Γκασίν Σνάιστερ. Απορρίπτω όμως την 130 και 131 γιατί διαγράφουν όλη την παράγραφο και δεν μας λένε τροπολογίες αυτές ποιες πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβάζονται και αυτό δημιουργεί ένα καθεστώς ασφάλειας. Όσον αφορά την τροπολογία 139 που διαγράφει την καταγραφή δεδομένων που προβλέπεται στην τροπολογία 116 τη μαγνητοσκόπηση, δεν μπορώ να υποστηρίξω την τροπολογία αυτή, γιατί μολονότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βίντεο, δεν έχουμε μαγνητοσκόπηση, ενδεχομένως να έχουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Σε περίπτωση που έχουμε μαγνητοσκόπηση, σε περίπτωση πτήσεων, θεωρώ ότι θα πρέπει αυτή να προστατεύεται από νομικής πλευράς. Για την 143 και 144 δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις τροπολογίες αυτές γιατί τα όσα προβλέπονται για την σωρό των θυμάτων δεν μπορούν να αποτελέσουν ποτέ αρμοδιότητα των αρχών ασφαλείας και διερεύνησης, είναι περισσότερο αρμοδιότητα των αστυνομικών αρχών και των δικαστικών αρχών. Θεωρώ λοιπόν δεν θα πρέπει να προβλέπονται τέτοιες διατάξεις για τις αρχές ασφάλειας. Πρέπει να σας πω ότι η Ισπανική Προεδρία τις τελευταίες αυτές εβδομάδες έχει δείξει ότι θέλει να καταλήξει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Προβλέπονται διάφορες συζητήσεις τριμερείς κατά τη διάρκεια του Ιουνίου και ελπίζω θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Βέβαια να σας πω ότι δεν θα, είναι, εύκολο το εγχείρημα για τα κράτη-μέλη ε, μένουν σε διάφορες θέσεις τους ιδίω όσον αφορά τις δικαστικές αρχές και από τη μία χώρα στην άλλη οι δικαστικές έρευνες αποκλίνουν πολύ. Τίθεται λοιπόν σταγματικό ζήτημα για ορισμένα κράτη-μέλη, τα οποία ενδεχομένως και να ήθελαν να περιορίσουν την ε, την πρόσβαση των δικαστικών αρχών στα εμπιστευτικά δεδομένα. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε όμως σε μια συμφωνία. Επίσης, σε πολλά κράτη-μέλη δεν είναι νόμιμο να κάνουν άλλες αρχές την έρευνα πέρα από τις δικαστικές αρχές το σημείο εκείνο που το Συμβούλιο ε, έχει μια ιδιαίτερα κλειστή θέση είναι για την αφορά των ε, συμβάντων, των δεδομένων. Το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου και ελπίζω τα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν κάπως την άποψή τους. Ελπίζουμε θα καταφέρουμε να τους πείσουμε ότι το να αναλύουμε τα συμβάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι καθοριστική σημασία προκειμένου να καταφέρουμε να αυξήσουμε το γενικότερο επίπεδο ασφάλειας και να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους επιβάτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Mr. Thank you, Mr. Chairman. I need to start by congratulating... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί πραγματικά έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Η στάση της ήταν πάρα πολύ επαγγελματική, δεν έχουμε σπουδαία πράγματα να προσθέσουμε. Πέντε τροπολογίες υποβάλαμε μόνο και ε, για τα υπόλοιπα σημεία συμφωνούμε και έχουμε και συμβαστικέ τροπολογίες βλέπω τώρα που, με τις οποίες συμφωνούμε. Έχουμε βέβαια μια επιφύλαξη και αυτή έχει να κάνει με το άρθρο 22 όπου αναφερόμαστε στα δεδομένα για τους συγγενείς των θυμάτων. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να φέρεται κυρίως σε συμβάντα, ατυχήματα και σε θέματα ασφάλειας. Ενώ εδώ πέρα βλέπουμε διατάξεις που αφορούν τελικά ένα άλλο ζήτημα, είναι λίγο εκτό θέματος. Και φοβάμαι ότι τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς. Αναφέρομαι στον κλάδο των αερομεταφορών που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά για να καλύψει άλλες ανάγκες, άλλους στόχους. Φοβόμαστε ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα τύχουν τη σωστή χρήση και γι' αυτό το λόγο έχουμε υποβάλει μια σχετική τροπολογία. Δεν συμφωνούμε με το άρθρο 22. Για όλα τα υπόλοιπα όμως όχι απλώς συμφωνούμε, τα βρίσκουμε καταπληκτικά και υποστηρίζουμε την εργασία που έχει κάνει η συγγήτρια. Κυρία Λίχτινγκ Ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Βεράκα για το ότι κατά τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων επέδειξε ανοιχτό πνεύμα. Ε, προσπάθησε λοιπόν τα διάφορα θέματα που συζητήσαμε να τα συμβιβάσει. Γνωρίζω ότι προέρχεται αντίδραση από το Συμβούλιο ε, και σε πάρα πολλά σημεία δεν κατανοώ γιατί εκφράζεται αυτή η αντίδραση. Βεβαίως υπάρχει το θέμα των ε, επικαλύψεων ε, στις ε, νομικές αναλύσεις, στις ποινικέ διώξεις πράξεων. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι πιστικό επιχείρημα για να υπάρχει τροποποιημένη και διαφοροποιημένη στρατηγική προλήψεων. Το Κοινοβούλιο λοιπόν οφείλει να μεριμνήσει για το πώς θα μπορέσουμε εμείς να περάσουμε τα αιτήματά μας. Μόνο αυτό σημαίνει πραγματική πρόληψη. Και αυτή την πρόληψη τη χρειαζόμαστε απόλυτα, καθότι αυτή τη στιγμή ασκείται τεράστια πίεση στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Στόχος μας είναι να αποφύγουμε ατυχήματα, άρα δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει και η βέλτιστη προστασία για τους αποκαλούμενους whistleblowers, για αυτούς ε, που μεταφέρουν ε, πληροφορίες από κύκλους οι οποίοι βρίσκονται κοντά κοντά στα συμβάντα. Αν δεν τους προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους θα παραμείνουμε και εμείς απλά σε επίπεδο θεωρίας και δεν θα υπάρχει καμία ουσιαστική πρόληψη. Θεωρώ λοιπόν ότι τα αιτήματά μας σε αυτόν τον τομέα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν αποδεκτά. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ από τους μεταρρυθμιστές συντηρητικούς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Δεβιράκ γιατί προγραμμάτισε και συνεδριάσεις εκτός των επίσημων συνεδριάσεων της Επιτροπής και την ευχαριστώ για το έργο της. Υπάρχει τεράστιος αριθμός τροπολογιών, δεν πρόκειται να τις σχολιάσω όλες. Θα επανέλθω σε ορισμένα σχόλια που είχα κάνει και στην αρχική συζήτηση. Εκεί που θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και έχω πολλέ επιφυλάξει είναι στο γεγονό ότι ο κανονισμό είναι τεχνικό και θα πρέπει να έχει τέτοια διατύπωση που να αναγνωρίζεται διεθνώ παρόλα αυτά, παρά τον τεχνικό του χαρακτήρα και τις εκτενείς συνεδριάς στην Επιτροπή, υπάρχει και μια πολιτική διάσταση στον κανονισμό αυτό, που είναι ευνόητη επίσης. Σε σχέση με το ζητούμενο, που είναι και η βελτίωση της επικοινωνίας με τους συγγενείς όταν σκέπτουν κάποια ατυχήματα, είναι αυτονόητο ότι θέλουμε καλύτερη ενημέρωση και θα πρέπει μεταφορείς, ε, οι οργανώσεις, οι εταιρείε να ενημερώνουν τους συγγενείς το συντομότερο δυνατό όταν έχουν τις πληροφορίες στη διάθεσή τους. Για το ρόλο της ΙΑΣΑ. Νομίζω ότι είπαμε ότι είναι πιστοποιητικός οργανισμός για τους ε, βιομήχανους και θα πρέπει να έχει κάποιο ρόλο συμβουλευτικό κατά προτίμηση. Κανένας δεν διαφωνεί με αυτό το στόχο. Κάτι άλλο που ανέκυψε και το συζητήσαμε, παρόλο που υπάρχει διάσταση απόψεων, αφορά την ε, δίκη, τη δικαστική διαδικασία και πώς λειτουργεί. Εμείς έχουμε ένα θεσμό που δεν ε, απαντάται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Κόρονερ, δεν υπάρχει υπετιότητα πολλές φορές και έτσι δεν πηγαίνει το, το ζήτημα στη δικαιοσύνη. Εμείς αντιμετωπίζουμε διαφορετικά το ρόλο της δικαιοσύνης, της δικαστικής εξουσίας και γι' αυτό θα πρέπει λόγω των διαφορών να προσέξουμε αυτό το θέμα. Τώρα, αν είναι ατύχημα ή συμβάν, αν ήταν τρομοκρατική απόπειρα ή αμέλεια, σίγουρα θα αναμειγνιόταν η δικαιοσύνη σε πρόωρο στάδιο, εφόσον υπήρχε ε, κατάφορη απόδειξη για το χαρακτήρα του ατυχήματος. Αλλά πολύ συχνά όταν έχουμε συμβάντη ατυχήματα, περνάνε χρόνια ολόκληρα για να διαλευκαθεί η υπόθεση. Μερικές φορές δεν διαλευκάνεται ποτέ. Και παρόλο που κατανοώ την πρόταση αυτή, θα πρέπει στη διατύπωση να είμαστε υπερβολικά σχολαστική και προσεκτική. Γενικώ είμαστε υπέρ μιας νοοτροπίας μη κατα, κατηγορίας και επαιτιότητας, γιατί αυτό κάναμε εδώ και 60 χρόνια στα περισσότερα ατυχήματα. Και αυτό συμβαίνει και διεθνώς με την ΙΚΑΟ. Δεν θέλουμε βέβαια παρέμβαση στο έργο των ερευνητών, γιατί χάρη στο δικό τους έργο σώθηκαν πολλέ ζωέ και ελπίζω να διασφαλιστεί ο υψηλό του επαγγελματισμό. Σε ό,τι αφορά τις ε, τροπολογίες, μια προφορική τροπολογία ε, ζητούσε περισσότερες πληροφορίες περί ασφάλειας των μεταφορέων. Αλλά καλύπτεται αυτή η απέτηση γιατί έχουμε και τη μαύρη λίστα στο μεταξύ. Υπάρχει υπάρχουν διαθέσιμε πληροφορίε δηλαδή. Και συμφωνώ εφόσον ε, γίνεται αυτό προς το συμφέρον των, του κοινού. Για το δίκτυο. Όλοι συμφωνούμε υπέρ του δικτύου και έχουμε τους καλύτερους επαγγελματίες του κόσμου που ασχολούνται με το θέμα αυτό στην Ευρώπη. Και αυτή την εμπειρογνωμοσύνη πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Είναι προφανές ότι είναι σωστό κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε για μια δημοσιονομική γραμμή. Όταν υπάρχει προϋπολογισμός, Φυσικά θέλουμε ένα κονδύλιο που θα επαρκεί για να υλοποιήσει το στόχο μας. Επίσης, ποιο είναι το πρόγραμμα εργασιών για το χρόνο. Θέλω ε, σωστή ενημέρωση και διεξοδική παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος και του προγράμματος εργασιών. Πώς θα λειτουργεί αυτό το δίκτυο. Δεν θέλουμε μια γραφειοκρατική δομή που θα επιβαρύνει τα πράγματα και δεν θα διορθώσει τίποτα. Αυτές τις διευκρινήσεις θα ήθελα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Τεβεϊράκ, ευχαριστώ και πάλι θερμά. Έχουν κανονιστεί πολλές τριμερείς συναντήσεις. Θα δούμε ποια θα είναι η έκβασή τους. Επίσης, ε, θα ήθελα να δω και ποια είναι η γνώμη του Συμβουλίου, γιατί πρόσφατα ακούσαμε πληροφορίες για πολύ θετική εξέλιξη στη θέση του Συμβουλίου. Δεν λέω ότι δεν χρειάζονται προσθήκες ή βελτιώσει από την Επιτροπή και δεν είμαι σίγουρη ότι τελείωσε η αναθεώρηση της αιτιολογικής σκέψης. Πάντως, ως προς το διατακτικό, η ομάδα μου συμφωνεί με την τελευταία εκδοχή της θέση του Συμβουλίου. Τώρα, για την ενημέρωση ως προς την εμφάνιση των συμβάντων, όχι τα ίδια τα συμβάντα. Επαναλαμβάνω, ο κανονισμός είναι τεχνικής υφής, οπότε αυτό το occurrence reporting την ενημέρωση της συχνότητας εμφάνισης μπορούμε να το ζητήσουμε ώστε να έχουμε όμως προαιρετική βάση και ο οικειοθελώς να γίνεται αυτή η ενημέρωση περί συχνότητας. Γιατί το 2002 είχαμε κάτι υποχρεωτικό αντίστοιχο στην Ευρώπη αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο που ακολουθήσαμε. Αυτά και περιμένω θετική έκβαση στο, στις τριμερείς συναντήσεις, ευχαριστώντας και πάλι την εισηγήτρια για την προσπάθειά της. Ευχαριστώ. Κύριος Δεγκράντες Πασκουάλ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ ειλικρινά και θερμότατα την εισηγήτρια Ντεβεϊράκ. Είναι πραγματικά η θέση της ε, πολύ ισορροπημένη και της εύχομαι καλή επιτυχία να φέρει σε αίσιο πέρας την έκθεσή της και μάλιστα πριν τελειώσει η Ισπανική Προεδρία. Εγώ έχω καταθέσει πέντε τροπολογίες συνολικά που θα μπορούσα να τις ανακεφαλαιώσω γύρω από δύο θέματα. Η πρώτη αφορά το εξή. Εδώ όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να δημοσιεύεται ο κατάλογος των θυμάτων. Το θέμα είναι πότε το γεγονός είναι αναφυσβήτητο. Και οι οικογένειες των θυμάτων δεν θέλουν μόνο να γνωρίζουν το κατά πόσο έχουν αναμειχθεί συγγενείς τους ε, στο ατύχημα, αλλά να υπάρχει μεμονωμένος εντοπισμός των, των θυμάτων. Και σήμερα υπάρχουν τεχνικά μέσα, ώστε χωρίς αμφιβολία χάρη στην εξέταση του DNA να ταυτοποιούνται όλα τα θύματα το συντομότερο δυνατόν. Και μάλιστα υπεράνω πάση αμφιβολίας για να γνωρίζουν οικογένειες. Στην Ισπανία είχαμε την καταδίκη ενός στρατηγού που εξαιτίας ε, αμέλειας ε, κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε παρά την καλή του πίστη και δυστυχώ θα δημιουργηθεί δικασμένο με αυτή την απόφαση. Ο άνθρωπο θα πάει στη φυλακή. Επίσης ε, υπάρχει ένα πρόβλημα ορισμών. Χρησιμοποιείται η όρος αιτία από την ΙΚΑΟ. Αλλά θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις των καιρών και να προσαρμοστούμε και εμείς στη νέα πραγματικότητα. Και οι πιλότοι και οι τεχνικοί και οι κυβερνήτες συμφωνούν όλοι στην διάκριση μεταξύ της τεχνικής έρευνας και της δικαστικής έρευνας. Η δικαστική έρευνα θα καταλήξει το κατά, κατά πόσο υπάρχει αστική ή ποινική ευθύνη. όρος όμως αιτία δεν είναι ουδέτερος. Είναι αποφασιστική σημασία και προδικάζει κάποιες συμπεριφορές. Οι Ιταλοί νομομαθείς θα θυμούνται την, ε, το παλιό δόγμα της αντικειμενικής ευθύνης. Βερσάρι είναι re όπως λέμε στα λατινικά. Τώρα, για την αιτία της αιτίας και για την αιτιολογική σχέση, αν χρησιμοποιήσουμε τον όρο αιτία, που δεν είναι ουδέτερος, παρόλο που λέμε ότι δεν προεξοφλεί η ποινική ή αστική ευθύνη, και μόνο η χρήση του όρου αιτία προδικάζει τέτοια ευθύνη. Και Μπορεί να έχουμε ε, την τεχνική έρευνα, αλλά μετά θα πρέπει η δικαστική εξουσία να κρίνει αν, υπήρχε, αν αιτία που να οδηγεί στην ε, επίρρηψη αστικών ή ποινικών ευθυνών. Χρησιμοποιώντας όμως ήδη από την τεχνική φάση της έρευνας τον όρο ευθύνη, κάουσα, τον όρο αιτία, κάουσα, προεξοφλούμε την ύπαρξη αστικής ή ποινική ευθύνης. Κάτι που είναι ένα μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό θα συμβεί. Ενώ δεν πρέπει να ισχύει κάτι τέτοιο, θα πρέπει η τεχνική έρευνα να προδικάζει τη δικαστική. Θα πρέπει να γίνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ των όρων ασφαλεία, των παραγόντων, παραγόντων ασφαλεία, τη τεχνική ευθύνη και τη ε, τεχνική έρευνα και των, α, της ανάλυσης που θα γίνει αργότερα στα πλαίσια της δικαστικής έρευνας ή της ανάκρισης. Και αυτή θα καταλήξει στο κατά πόσο υπάρχει αστική ή ποινική ευθύνη. Και η ίδια η ΚΑΟ θα πρέπει να τροποποιήσει την ορολογία που χρησιμοποιεί. Γιατί η νομολογία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν όλα αυτά για να δοθούν τα εχέγγυα στα θύματα, στους κατηγορούμενους αλλά και στις οικογένειες. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ήδη από την αρχή όρος αιτία γιατί θα είναι τεράστιες συνέπειες που θα έχει η χρήση αυτού του όρου και για τη μεταγενέστερη δικαστική διαλεύκαση της υπόθεσης. Ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ θερμά την εισηγήτρια για το έργο της και να πω ότι υπάρχουν τρία σημεία στα οποία επιμείναμε και συμπεριλήθηκα στην έκθεση. Καταρχήν σε ό,τι αφορά τα θύματα, νομίζω ότι είναι μεγάλη ευαισθησία που έδειξε ε, η συγγετρία, αλλά χρειάζεται και επαγγελματισμό. Ευαισθησία για τη συμπαράσταση προ τα θύματα και ενημέρωση, αλλά και επαγγελματισμό που απαιτείται από την αρχή για να δοθούν αξιόπιστες πληροφορίες. Η αξιοπιστία των πληροφοριών είναι σημείο κέρια σημασίας. Το θέμα δεν θα είναι πότε θα δημοσιευθεί ο κατάλογος με τα θύματα σε μισή, μία ή δύο ώρες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι πληροφορίες να είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Και σίγουρα δεν θα πρέπει να υπερέχουν εδώ οικονομικά κριτήρια, κριτήρια ανταγωνισμού. Εδώ αυτό που προέχει είναι να διχθεί μια ανθρωπιά απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων. Επίσης, ό,τι αφορά τη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και τη δικαστική έρευνα, θα πρέπει καταρχήν να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία όλων όσων προσπαθούν να βρουν λύσεις κάνοντας μια τεχνική ανάλυση και έρευνα. Είναι σαφής ο ρόλος τους και ο ρόλος της δικαιοσύνης έρχεται σε δεύτερη φάση. Με επίσης διαφύλαξη της ανεξαρτησίας φυσικά της δικαστικής έρευνας. Αλλά νομίζω ότι το κείμενο τα διασφαλίζει όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά την τεχνική, θα πρέπει φυσικά να προσαρμόζεται σε ένα διεθνές πλαίσιο, προβλέποντας τη δυνατότητα και αναθεώρησης είτε ευρωπαϊκής είτε ε, διεθνούς. Γιατί και τα διεθνή κείμενα μπορούν στο μέλλον να αναθεωρηθούν. Επειδή υπάρχει μια διεθνή συμφωνία δεν σημαίνει σαν και κολλά ότι είναι αμετακίνητη ή δεν επιδέχεται αλλαγών. Πάντως η προσέγγιση είναι σωστή ότι υπάρχουσες σε συνθηκες συμβάσεις και οι συνεργασίες ε, μπορεί ενδεχομένως να τύχουν και Επίσης, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και στην πρόληψη. Να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Γιατί αν τα συμπεράσματα ενός αεροπορικού ατυχήματος δεν οδηγήσουν σε μια βελτίωση της κατάστασης, σε βελτίωση και τεχνικής υφής, τότε θα είναι πραγματικά κρίμα. Βέβαια, μερικές φορές υπάρχει μία νοσηρή εισήχηση, ένα μπέρδεμα μεταξύ της ε, εμπλεκόμενης αεροπορικής εταιρείας και του εμπειρογνώμονα που κάνει τεχνική έρευνα. Μερικές φορές υπάρχει μπέρδεμα και στη δικαιοσύνη. Τέτοιες συγχύσεις θα πρέπει να τις αποφύγουμε. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του ατυχήματος, μερικές φορές συγκροτούνται και ad hoc κοινοβουλευτικές επιτροπές που επικεντρώνονται όμως στο πολιτικό επίπεδο, σε πολιτική συζήτηση και αμελούν το τεχνικό, κάτι που οδηγεί σε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση της διαλεύκανσης της έρευνας. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν και τα δικαιώματα της δικαιοσύνης, αλλά και την ευαισθησία και την συμπαράσταση προς οικογένειες των θυμάτων. Ευχαριστώ. Ο Σαΐδελ Καντράουι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα το συγγνώμη, έφτασα καθυστερημένο και έχασα την παρουσίαση που έγινε στην αρχή. Ο Σιώδη ηγητή μα δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μα. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα μπορούσε να τύχει γενικότερη συμφωνία. Ξέρουμε ποιε είναι οι προτεραιότητε, οι βασικέ. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι με τι προτεραιότητε αυτέ και τα όσα είπε ο κύριο Γκρό επίση είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τη δική μα την ομάδα. Το σημαντικό είναι οι έρευνες να γίνονται με τρόπο αποτελεσματικό, να οδηγούν σε καλά αποτελέσματα. Και είναι σημαντικό να έχουμε πλέον και μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για τις έρευνες αυτές. Και αυτό θα πρέπει να γίνει, έχοντας βέβαια κατά νου το ότι ε, και η ε, δικαστική εξουσία θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις ευαίσθητες πληροφορίες, στα εμπιστευτικά δεδομένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει όμως να λυγίσουμε απέναντι στις πιέσεις που ασκούν τα κράτη-μέλη. Τα πράγματα θα πρέπει να διευθετηθούν με σωστό τρόπο. Όσον αφορά τώρα τη βάση δεδομένων. Και αυτή θα πρέπει να συνάδει με τα κριτήρια τα οποία, τα οποία εμείς θέλουμε. Θέλουμε μια βάση δεδομένων με ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Νομίζω ότι μπορούμε όλες να συμφωνήσουμε σε αυτό. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι συμφωνούμε τα περισσότερα σημεία. Σας ευχαριστούμε κύριε Μάσερ. Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να πω τίποτα σπουδαίο. Κατ' ουσίαν οι συνάδελφοι προαλήσαντες με κάλυψαν. Εγώ θέλω μόνο να υπογραμμίσω ότι κατά τη δική μας άποψη είναι καθοριστική σημασία να δει κανεί ε, αυτά τα ατυχήματα που προκαλούνται στην ε, πολιτική αεροπορία. Θα πρέπει να ερευνηθούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποφευθούν την επόμενη φορά ή δυνατόν. Αυτό είναι το θέμα που μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να προχωρήσουμε με ευαισθησία και να δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτούς που γνωρίζουν κάτι να το πούν χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο να καταστούν ύποπτοι. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα πρέπει να διευκρινιστεί από τι προκλήθηκε το ατύχημα και μετά το θέμα είναι να δει κανεί ε, ποιος ε, φταίει. Είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο θέματα γιατί τελείως δεν θα προχωρήσουμε. Η εισηγήτρια Σωστά λοιπόν το ίδιο το θέμα και γι' αυτό και εμείς ε, υποστηρίζουμε την εκθεσή της. Ε, το μόνο αυτό το 22 ε, το είπε ο συνάδελφος και διαφέρει λιγάκι απόψή μας λόγω της προστασίας των δεδομένων αλλά κατά τα άλλα θεωρούμε ότι σωστή είναι η προσέγγιση γιατί στόχος μας είναι να αποφευθούν οι δυνατόν στο μέλλον ατυχήματα στις αεροπορικές μεταφορές. Πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν, θα ήθελα να πω και εγώ μερικά λόγια. Κοιτάξτε, όταν ξεκινήσαμε νομίζω ότι υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά στην ε, ανεξαρτησία των ε, ερευνών ε, που λαμβάνουν χώρα. Και επίσης αυτό που μας ενδιαφέρει ήταν και ποιος ήταν ο ρόλος της, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας στα πλαίσια των ε, ερευνών. Αυτό λοιπόν που ενδιαφέρει είναι, όπως είπαμε πολύ σωστά, να παραμείνει η ανεξαρτησία των ε, ερευνητών και να υπάρχει και ο ρόλος εκείνου που αναλαμβάνει την διερεύνηση της υπόθεσης Σύμφωνα με τον ΙΚΑΟ δεν μπορεί κανείς να είναι και ρυθμιστής και ε, ερευνητής της υπόθεσης και να ερευνά την υπόθεση. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Αφορά στο θέμα του χρονικού διαστήματος δηλαδή στην ενημέρωση των συγγενών των θυμάτων σε περίπτωση ατυχήματος. Εγώ συμφωνώ εδώ με αυτά που είπε ο κύριος Γκρός. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να υπάρχει ο ακριβής κατάλογος των θυμάτων και όχι ένας πρόχειρος και προσωρινός που μπορεί να είναι και λανθασμένος. πολλοί ζητούν ο ακριβής αυτός κατάλογος να καταρτιστεί μέσα σε 30 λεπτά. Εγώ λοιπόν προτείνω το να προτείνουμε το κατάλογο αυτό ε, στη διάρκεια μέσα σε μιας ώρας. Αυτό είναι ε, δικλείδα ασφαλείας γιατί με τον τρόπο αυτό πράγματι δεν διατρέχουμε κίνδυνο να δώσουμε λάθος πληροφορίες όταν υπάρχει και μια τέτοια τραγική κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα να σκεφτείτε ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο κατάλογος δεν είναι σωστός και όχι να συνταχθεί το συντομότερο δυνατόν. Βεβαίως, μέσα σε... στα δελτία ειδήσεων, οι άνθρωποι των δελτίων ε, θέλουν τον ακριβή κατάλογο ή δυνατόν εχθές. Και γι' αυτό κατανοώ ότι αν ε, χρειαστούμε άπλετο χρόνο για να ε, ενημερώσουμε τους ε, συγκινήσεων των θυμάτων, τότε ξέρετε τι θα γίνει. Έτσι και αλλιώ θα ενημερωθούν από τα δελτία ειδήσεων. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι οι δύο ώρες είναι ικανοποιητικό χρονικό διάστημα. Προσφέρει τη δυνατότητα να καταρτήσει κανείς έναν ακριβή κατάλογο χωρίς λάθη και αυτό που έχει καθοριστική σημασία για μένα, όπως σας λέω, είναι ο κατάλογος αυτός να είναι ακριβής. Και θεωρώ ότι εάν πέσουμε κάτω από αυτό το χρονικό διάστημα, ελοχεύει ο κίνδυνος να γίνουν λάθη είτε διότι οι αεροπορικές εταιρείε ε, είναι υποποίηση, είτε διότι ασκούν πίεση οι ίδιοι οι συγγενείς. Το τρίτο θέμα που θέλω να θίξω αφορά στην ε, πρώτη ανάγνωση ή οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό. Ε, Βεβαίω ε, κατανοώ ότι η Ισπανική Προεδρία θέλει να τα περάσει όλα τα θέματα που χειρίζεται στην πρώτη ανάγνωση. Όμω, ξέρετε, υπάρχουν και περιπτώσει που πρέπει λιγάκι να του συγκρατήσουμε και να του πούμε ότι υπάρχει εδώ και ένα κοινοβούλιο και προβλέπεται ρόλο για το κοινοβούλιο. Σε κάποια σημαντικά θέματα σε αυτή την έκθεση εξακολουθεί να υφίσταται διάσταση απόψεων ανάμεσα στο κοινοβούλιο και το συμβούλιο. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση η συγγήτρια να συνεχίσει να δούμε τι θα γίνει αύριο στην ψηφοφορία και στην Ολομέλεια και με τον τρόπο αυτό να καταλήξει μια συμφωνία με την Ισπανική Προεδρία. Όμως συνιστώ σύνεση στο να υπάρχει πάση θυσία ε, απόφαση κατά την πρώτη ανάγνωση τη στιγμή που όπως σας είπα υφίστανται διαφορές όσον αφορά ε, την διερεύνηση μιας υπόθεσης ε, που ακριβώς επιλαμβάνει του θέματος ε, η δικαστική εξουσία. Βλέπετε αυτό είναι ένα καθοριστικό θέμα όπου υπάρχει διάσταση απόψεων. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε μια καλή νομοθετική πράξη και όχι κάτι που να βολεύει την Ισπανική Προεδρία μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ε, θα έλεγα λοιπόν, βεβαίως ε, και δέχομαι αυτά που λέει η συγγήτρια, παρόλα αυτά να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί. Δεν θέλω να ε, αποσπάσω την προσοχή σας από αυτό που κάνετε, να διαπραγματευτείτε με το Συμβούλιο ε, και με βάση αυτά που θα αποφασίσει το Κοινοβούλιο αύριο και στην Ολομέλεια. Έτσι λοιπόν, εκ μέρου τη ε, Κομισιόν, ο κύριο Χέρκε. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Σίμψον. Θα ήθελα καταρχά να συγχαρώ την κυρία Ντεβέρακ για την πολύ σκληρή δουλειά που έκανε, την καταπληκτική της δουλειά στο ζήτημα αυτό πάντα είμαστε συνηθισμένοι στο να έχουμε καταπληκτικέ εκθέσει από την κυρία Ντεβέρα και για παράδειγμα μπορώ να αφαιρθώ στην νομοθεσία για την ε, μαύρη λίστα. Επομένω και στην περίπτωση αυτή θα θέλω να ευχαριστήσω για την πολύ καλή δουλειά τη. Έχετε πραγματικά εντοπίσει πολύ καλά τα βασικά ζητήματα και η συζήτηση δείχνει ότι έχετε συνειδητοποιήσει ποια είναι τα βασικά ζητήματα και βλέπω ότι υπάρχει ένα μεγάλο βαθμό σύγκληση ανάμεσα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φαίνεται ότι όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε να εξυγχρονίσουμε το υφιστάμενο νομοθετικό σύστημα, θέλουμε να ενδυναμώσουμε το νομοθετικό αυτό σύστημα και θέλουμε να ενισχύσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τους κανόνες που υφίστανται στον τομέα αυτό, προκειμένου να μας σε θέση να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά την ασφάλεια. Πολλοί Βουλευτέ, το είπαν ότι πρέπει να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τα ατυχήματα προκειμένου να τα προλάβουμε αυτά στο μέλλον, να μην συμβούν στο μέλλον. Και αυτό βρίσκεται πραγματικά πίσω από τη βασική ιδέα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε μια οδηγία στο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει τώρα ένα κανονισμό, δηλαδή ένα νομοθετικό σύστημα πολύ πιο ισχυρό. Για τα διάφορα ζητήματα τα οποία έθιξαν οι βουλευτέ θα είμαι πολύ σύντομο και θα απαντήσω στις, στα σχόλιά σα. Καταρχά, όσον αφορά το δίκτυο των αρχών διερεύνηση έχουμε τις ανεξάρτητες αρχές, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει εδώ πέρα να δημιουργηθεί ένα δίκτυο αρχών διερεύνησης και συμφωνούμε την κυρία Ντεβέιρακ ότι ε, θα πρέπει το δίκτυο αυτό να αποτελέσει ένα σώμα συντονισμού, να μην λειτουργεί απλώς σε εθελούσια βάση όπου ενδεχομένως να συζητάνε ατύπως οι αρχές διερεύνησης. Χρειαζόμαστε κάτι πιο ισχυρό. Θέλουμε ένα δίκτυο το οποίο να έχει μια ισχυρή εντολή, να μπορεί να λαμβάνει δράση και να αποτελεί προστιθέμενη αξία για την ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δίκτυο αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει και τα μικρότερα κράτη-μέλη που δεν έχουν του απαραίτητου πόρου να δημιουργήσουν αρχέ διερεύνηση. Γι' αυτό το λόγο είμαστε υπέρ των τροπολογιών εκείνων που θέλουν καλύτερο ορισμό της αποστολής του δικτύου αυτού και θέλουμε και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα ετήσιο επίσημο πρόγραμμα εργασίας. Δεν προτείνουμε εδώ πέρα να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε εδώ πέρα μια δομή πιο ελαφριά. Η κυρία Φώστερ υπέβαλε δύο ερωτήματα. Πρώτον για τον προπολογισμό. Στο δημοσιονομικό δελτίο προβλέπονται 0,6 εκατομμύρια ευρώ για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Θεωρούμε ότι αρκούν οι πόροι αυτοί και τι θα κάνει βέβαια το δίκτυο αυτό. Θα λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντολές προκειμένου να προτιμάζει μηχανισμούς για ανταλλαγή πληροφοριών και πόρων, για συντονισμό της κατάρτισης, για ανάλυση των συστάσεων ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για την παροχή συμβουλών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιμένουμε όμως ότι δεν πρόκειται για έναν νέο οργανισμό, μιλάμε για μία επισημοποίηση ενός μιας άτυπης συνεργασίας αρχών διερεύνησης που ήδη φίσταται ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Το δίκτυο αυτό αρχών διερεύνησης δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τις εθνικές αρχές διερεύνησης. Δεύτερον, πολλά ερωτήματα αναφέρθηκαν για το σύστημα υποβολής αναφορών. Η κυρία Ντεβέιρακ νομίζω ότι έχει υιοθετήσει τη σωστή προσέγγιση. Οι τροπολογίες συμπληρώνουν και επεκτείνουν περισσότερο τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε καλύτερη χρήση των πληροφοριών που έχουμε για τη συχνότητα εμφάνιση συμβάντων στον αεροπορικό τομέα και θέλουμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί με αυτόν τον τρόπο όσον αφορά την πρόληψη των ατυχημάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσέγγιση αυτή είναι πολύ σημαντική και θα μας επιτρέψει να σημειώσουμε πρόοδο στο μέλλον. Στον κανονισμό αυτό θα πρέπει να διευθετηθούν όλα αυτά και όχι αργότερα. Τώρα θα πρέπει να διευθετήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα, όσον αφορά το ρόλο τη ε, ΕΑΖΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλεια Αεροπορία, νομίζω ότι ο κύριο Σίμψον εξήγησε τα πράγματα πολύ καλά. Θέλουμε ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια Αεροπορία να έχει συμβουλευτικό ρόλο. Θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμό ανάμεσα στον καονισμό και την έρευνα των ε, ατυχημάτων. Δεν είναι ρόλο τη ΕΑΖΑ να ερευνεί τα ατυχήματα. Πάντω θα πρέπει η ΕΑΖΑ να έχει πρόσβαση στι πληροφορίε γιατί ως αρχή υπεύθυνη για την πιστοποίηση των αεροσκαφών είναι πολύ σημαντικό να έχει και αυτή τις πληροφορίες αυτές για να αντιμετωπίζει προβλήματα ασφάλειας τα οποία εντοπίζουν οι αρχές ασφάλειας και οι αρχές έρευνας. Σαφώς όμως θα πρέπει να καθορίσουμε σαφώς τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της ΕΑΖΑ, γιατί όταν συμβαίνει ένα ατύχημα δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου για να προσπαθούμε εκείνη τη στιγμή να δούμε ποιος κάνει τι όσον αφορά τα θύματα και τον κατάλογο. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ ευαίσθητο και υπάρχουν και κάποια νομικά ζητήματα βέβαια σχετικά με το ζήτημα αυτό. Το Συμβούλιο εν γέννη είναι υπέρ της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή το συντομότερο δυνατό, το αργότερο μέσα σε δύο ώρες λέγεται, στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την προθεσμία. Σαφώς όλοι είμαστε υπέρ της ε, πιο σύντομης εφικτής προθεσμίας. Θεωρούμε ότι έχουμε τα τεχνικά μέσα για να καταλήγουμε στον κατάλογο αυτό πάρα πολύ γρήγορα σήμερα. Ενδεχομένως να είναι δύσκολο να επιβάλλουμε βέβαια τις υποχρεώσεις αυτές σε τρίτες χώρες, σε αεροδρόμια τρίτων χωρών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Σίμψον. Πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς και να είμαστε απόλυτα ακριβείς στον κατάλογο αυτό. Θέλουμε έναν ακριβή κατάλογο το συντομότερο δυνατό, αφού είναι το ευκταίο και θεωρώ ότι η προθεσμία των δύο ώρων να είναι ενδεχομένως η καλύτερη δυνατή συμβαστική λύση και θα πρέπει αυτό να συνδυαστεί με την ανάγκη της απαραίτητης παροχής βοήθειας προς τις οικογένειες των θυμάτων. Και γι' αυτό τον λόγο προτείνουμε σε εθνικό επίπεδο να υπάρχουν αρχές που να ασχολούνται με το σημαντικό αυτό ζήτημα. Τελευταίο τώρα σημείο. Η σχέση ανάμεσα στην έρευνα τη ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Και για το σημείο αυτό θεωρώ ότι Μάλλον στο σημείο αυτό έχουμε, αν θέλετε, και τις μεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά τη διαδικασία συνδιαλλαγής, όσον αφορά την έβρεση συμβιβασμού. Υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα, αναφέρθηκε η κυρία Φώστερ σε αυτό, ο κυρίος Ντεγκράντες Πασκουάλ επίσης αναφέρθηκε στο σημείο αυτό με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Εμείς θεωρούμε ότι ο μόνος στόχος της έρευνας των ατυχημάτων θα πρέπει να είναι η πρόληψη των ατυχημάτων και δεν είναι στόχος της έρευνας να επιρρύπτει την ευθύνη. Η έρευνα των ατυχημάτων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να χωριστεί από τις υπόλοιπες δικαστικές έρευνες. Έχουμε όμως μια βασική δυσκολία και αυτή έχει να κάνει με τις διαφορές που υπάρχουν στο Σύνταγμα των κρατών μελών. Σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι οι δικαστικές αρχές αυτές οι οποίες αναλαμβάνουν τον έλεγχο της έρευνας και έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε στοιχεία θέλουν για την ε, ανάλυση της κατάστασης και για να καταλήξουν σε μια δικαστική απόφαση. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν, δεδομένου των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη, να διαχωρίσουμε την εξουσία ανάμεσα στη δικαστική εξουσία ουσιαστικά και την εξουσία που έχει η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Μπορούμε να αποδεχτούμε βέβαια τους συνταγματικούς περιορισμούς που υπάρχουν και παράλληλα να δώσουμε όλα τα απαραίτητα μέσα στους διερευνητές ώστε να μπορούν τουλάχιστον να επιτελέσουν σωστά την τεχνική τους ανάλυση και να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα αυτά τα μέσα τα οποία χρειάζονται προκειμένου να είναι σε θέση εξ αρχής να δούνε τι ακριβώς έγινε. Και θα πρέπει για αυτό το λόγο να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν και μεταξύ τους πληροφορίες από τη μία χώρα στην άλλη. Καταλαβαίνω ότι αυτό το σημείο θα είναι το πιο δύσκολο στα πλαίσια της ε, συνδιαλλαγής. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προχωρήσει και αυτή γρήγορα. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα συναντήσουμε δυσκολίες. Επίσης πιέζει το χρονοδιάγραμμα. Ας κάνουμε τουλάχιστον την προσπάθεια και θα δούμε πώς θα πάμε. Όπως είπε και ο κύριος Σίμψον, πιστεύουμε και εμείς ότι θα πρέπει να έχουμε τελικά μια καλή νομοθεσία, ότι σε αυτό θα πρέπει να στοχεύουμε, όπως σας είπα, για πάρα πολλά σημεία υπάρχει ήδη μια σημαντική σύγκληση, ενδεχομένως να υπάρξουν περισσότερες δυσκολίες σε κάποια σημεία, αλλά νομίζω θα πρέπει να αφήσουμε τη δικασία της συναπόφασης να τρέξει και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε στο τέλος να καταλήξουμε σε μια καλή νομοθεσία. Και αν, δεν τα πετύχουμε στα πλαίσια, αν το πετύχουμε στα πλαίσια της Ισπανικής Προεδρίας, τόσο το καλύτερο, γιατί θα καταφέρουμε ε, πολύ γρηγορότερα να ενισχύσουμε το εφιστάμενο σύστημα ασφάλεια. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κυρία Ντεβέρα και έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη διαμόρφωση της έκθεσης αυτής, τη βελτίωσαν και σε τελική ανάλυση καταλήξαμε σε συμφωνία για πολλά σημεία. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που είπαν ο κύριος Κασίν και η κυρία Μάισνερ για τα στοιχεία προς τους συγγενείς. Δείτε την τροπολογία 56 που δίνει εχέγγυα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κυρία Λίχτεμπέργκερ, μιλήσατε για την ανάγκη ε, υπεροχής της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Καλά, δεν πειράζει. Αργότερα. Η κυρία Φώστερ μίλησε για τη σχέση μεταξύ της τεχνικής έρευνας, ε, της έρευνας ασφάλειας και της δικαστικής έρευνας. Όντω, αυτό είναι το πιο λεπτό σημείο τη έκθεση. Και γι' αυτό θα πρέπει να θεσπίσουμε κανόνε που θα προβλέπουμε σαφήνεια τι μπορεί να διανεμηθεί στη δικαιοσύνη, τι θα διαβιβαστεί και τι θα μείνει ε, απόρριτο. Γι' αυτό έχουμε και την τροπολογία 40. Αλλά σίγουρα οι ένομε τάξει ενδιαφέρουν στο σημείο αυτό και στην αντιμετώπιση που υιοθετούν. Η κυρία Φώστερ μίλησε για το δίκτυο, τη θέσπιση του δικτύου. Απάντησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σημείο αυτό. Όταν υπέβαλα το σχέδιο εργασία, το έγγραφο εργασία, είπα ότι σε καμία περίπτωση αυτό το δίκτυο δεν θα γίνει ένα νέο στρώμα γραφειοκρατία, μια νέα γραφειοκρατική δομή. Απλώ θα διευκολύνει τα γραφεία με τις χαμηλότερες επιδόσεις ε, να κερδίσουν το χαμένο έδαφος. Μιλήσατε, κυρία Δεγκράντες, για τον ορισμό της ΟΑΣΕΑ. Αλλά το θέμα αυτό δεν είναι δικό μας θέμα, γιατί αλλού λαμβάνονται αποφάσεις για τους ορισμούς αυτούς. Η κυρία Λίχτεμπέργκερ, κύριε Πρόεδρε, μίλησε για την ανάγκη υπεροχή τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σα καθησυχάσω, επουδενή δεν θα εκποιήσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να καταλήξουμε πάση θυσία σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Φυσικά θα δώσουμε τη μάχη στις διαπραγματεύσεις, αλλά εμένοντας στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εσείς κύριε Πρόεδρε και κύριος Γκρός μιλήσατε για την ανάγκη αξιόπιστων πληροφοριών. Χρειαζόμαστε φυσικά ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες. Αλλά και το στοιχείο χρόνος είναι σημαντικό. Γιατί οι οικογένειες αγωνιούν αν κάποιος συγγενής τους έχει εμπλέκει στο δυστύχημα αυτό το αεροπορικό. Πήγαμε στο αεροδρόμιο του Ζάβεντεμ στις Βρυξέλλες και διαπιστώσαμε ειδήσει όμως ότι μέσα σε μία ώρα μπορεί να, εκδοθεί ένα, να δημοσιευθεί ένας αξιόπιστος κατάλογος. Εδώ δεν θα κάνουμε παζάρια αν θα δημοσιευθεί ο πίνακα σε μισή μία ώρα. Βέβαια, ο χρόνος περνάει πολύ αργά για τις οικογένειες που αγωνιούν και περιμένουν πώς και πώς να μάθουν αν ο συγγενής τους βρισκόταν στο αεροπλάνο. Επίσης, κύριε Γκρός, είναι σημαντική σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ανάλυση των στοιχείων του ΕΚΕΡ. Ο Σαΐντελ Καντράου είπε ότι θα πρέπει να εμείνουμε πιστοί στην αρχή του διαχωρισμού μεταξύ της τεχνικής έρευνας, της έρευνας ε, για την ασφάλεια και της δικαστικής έρευνας. Συμφωνώ και εγώ με την ανάγκη σαφούς διαχωρισμού. Αυτά νομίζω ότι σχολίασα σχεδόν όλες τις παρατηρήσεις. Σας ευχαριστούμε κυρία Ντεβεϊράκ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στην Επιτροπή μας για την έκθεση αυτή και θα περάσει την Ολομέλεια είτε του Ιουλίου είτε του Σεπτεμβρίου αλλά ακόμη δεν είναι βέβαιο σε ποια από τι δύο. Πάντως μετά την αυριανή ψηφοφορία θα έχετε ευκαιρία να συνεννοηθείτε με τους σκιώδεις συγκητές σα για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Εντάξει, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που κανονικά είναι η γνωμοδότηση Βλάσακ για τον καθορισμό προτύπων για τις επιδόσεις των καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων αλλά ο κύριο Βλάσακα αναμένεται στην αίθουσα μετά από ένα τέταρτο 20 λεπτά. Θα έλεγα λοιπόν να περάσουμε μια και ο συντάκτης Αλκαντράουι είναι παρόν, να εξετάσουμε τη δική του γνωμοδότηση. Μάθιου, δεν πας να βρεις τον κύριο Κούν που είναι και σκιώδης. Αν δεν έχει αντίρρηση να εξετάσουμε τώρα τη γνωμοδότησή του κύριου Αλκαντράουι, θα μας βοηθήσει πολύ. Εντάξει, Σαΐντ. Ωραία. Πρόκειται για τον έλεγχο από τα κράτη-μέλη τη άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Σημείο 8. Σαντ, έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εδώ πρόκειται για θέματα προπολογισμού. Υπάρχουν πολλοί που δεν του αρέσει το θέμα αυτό, αλλά είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε γιατί ε, ασκεί επιρροή στι αποφάσει μα και όχι μόνο ε, το θέμα της ε, θέσπης νόμων αλλά και εφαρμογή τους και αυτό είναι καθοριστική σημασία. Να πω λοιπόν κάτι για την ιστορία του θέματος. Ησυχία παρακαλώ λέει ο πρόεδρος, αν έχετε καλοσύνη ε, ησυχία στην αίθουσα. Αν θέλετε να έχετε ιδιωτικές συζητήσεις παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι τις συζητήσεις αυτές να τις κάνετε έξω και αν έχετε καλοσύνη να βγείτε σιγά, χωρίς θόρυβο, έξω από την αίθουσα. Λοιπόν, να πω κάτι για την ιστορία του θέματος. Μέχρι πριν από λίγο καιρό είχαμε τη διαδικασία της ε, επιτροπολογίας. Κατά κάποιον τρόπο αυτή ήταν μια διαδικασία ελέγχου. Εκεί είχαμε το δικαίωμα να καταθέσουμε βέτο κάτω από ορισμένες ε, προϋποθέσεις. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι ήμασταν σε θέση να εκφράσουμε αντιρρήσεις οποτεδήποτε η Κομισιόν υπερέβαινε τις αρμοδιότητες της. Ε, ε, κατόπιν υπήρχε και η διαδικασία της συναπόφασης ε, για σημαντικά θέματα. Τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχουν δύο διαδικασίες που έχουν απομείνει. Είναι δύο σημαντικές διαδικασίες, όπως ξέρετε όλοι, η παλιά διαδικασία της επιτροπολογίας τώρα πλέον μετατρέπεται είτε στα Delegated Acts, Και αυτό είναι κατά κάποιον τρόπο αυτό που αποκαλούμε ε, σήμερα ε, πράξεις κατεξουσιοδότηση. Παράλληλα με τις ε, πράξεις κατεξουσιοδότηση υπάρχουν και οι εκτελεστικές πράξεις. Ε, πρόκειται για το άρθρο 91 και ε, το Κοινοβούλιο προετοιμάζει μία τοποθέτηση, μία γνωμοδότηση προς την Νομική Επιτροπή. Το καθοριστική σημασία θέμα είναι τώρα το εξής πότε έχουμε να κάνουμε με πράξη κατεξοδότηση και πότε με εκτελεστική πράξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να μην χρειαστεί κάθε φορά να συζητάμε εκ νέου για το θέμα αυτό. Η συζήτηση λοιπόν είναι καθοριστική σημασία κυρίως για τις επιτροπές εκείνες όπου η διαδικασία της συναπόφαση είναι καινούρια όπω Γεωργική Επιτροπή, ε, Εμπορική Επιτροπή πάνω στο θέμα είναι το εξή. Παλαιότερα υπήρχαν θέματα που δεν υπόκειντο στη διαδικασία του ελέγχου. Ε, τώρα όμως υπάρχουν πλέον σε κάποιο έλεγχο και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ στην ουσία εκθεσή μου. Εμένα με ενδιαφέρουν κατά κύριο λόγο δύο πράγματα. Πρώτον, η πρόσβαση στις πληροφορίε. Αυτό για μένα είναι καθοριστική ε, σημασίας. Η Κομισιόν αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παραθέτω ε, το Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να ενημερώνεται... στα τακτά χρονικά διαστήματα τέλος παράθεσης σχετικά με τις αποφάσεις των αρμόδιων επιτροπών. Ίσως ε, να γνωρίζετε ότι υπάρχει μια ολόκληρη σειρά προτάσεων που αφορά ε, στις ε, εκτελεστικές πράξεις. Εμένα με ενδιαφέρει το ότι ε, τις πληροφορίες αυτές πρέπει να τις παίρνουμε παράλληλα με τα κράτη-μέλη. Δηλαδή ε, θα πρέπει να ε, βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο με τα κράτη-μέλη. Σήμερα όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο με τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Και επίσης θεωρώ ότι ως παρατηρητές θα πρέπει να μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις επιτροπές. Εξάλλου δεν ισχυρίζομαι ότι πρέπει πάση θυσία να κάνουμε χρήση αυτού του θέματος. Ε, Πάνω στα πρέπει να είναι δυνατό. Και ε, επίσης ε, μπορούμε να στείλουμε και έναν υπάλληλο ο οποίος να ενημερώνεται άμεσα. Άρα δηλαδή εγώ δεν ζητώ περισσότερες αρμοδιότητες, απλά ζητώ να υπάρχει ενίσχυση της ενημέρωσης ε, προς την ε, κατεύθυνση του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι καλύτερο για τη διαφάνεια και έτσι λοιπόν είμαστε και καλύτερα σε θέση να διαπιστώσουμε κατά πόσο η Επιτροπή ενδεχομένω υπερβαίνει τις ε, αρμοδιότητές της. Εδώ λοιπόν ε, προκύπτουν κάποιες δυσκολίες, οι οποίες και εγώ εξετάζω στην έκθεσή μου. Η διαδικασία είναι η μετάβαση από την τρέχουσα διαδικασία στη διαδικασία μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Εμείς ε, καλούμε την Κομισιόν το σύνολο της ε, νομοθεσίας, οπουδήποτε εμφανίζεται η έκφραση επιτροπολογία, να προσαρμόσει το κείμενο ε, στην ε, νέα ορολογία και μάλιστα να εξετάσει όλες ε, τις ομοθετικές πράξεις που υπάρχουν σε σχέση με την Επιτροπολογία για να διαπιστωθεί ποιες είναι οι νέες διαδικασίες που ισχύουν τώρα. Η Κομισιόν εξάλλου πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον ε, πρόκειται για πράξη κατά εξουσιοδότηση ή Η πρόταση της Επιτροπής δεν είναι αρκετά προχωρημένη. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι ο έλεγχος παραμένει ως είχε στο παρελθόν και οι άλλες διαδικασίες τις οποίες σας παρουσίασα προηγουμένως θα αντικατασταθούν από τις εκτελεστικές πράξεις τις οποίες δεν μπορούμε να επηρεάσουμε στον ίδιο βαθμό. Ε, σας λέω λοιπόν ότι δεν μπορούμε αυτές τις τέσσερις παλιές κατηγορίες να τις εντάξουμε όλες σε μία νέα κατηγορία ε, δεν μπορούμε όλα αυτά να τα εντάξουμε στις εκτελεστικές πράξεις. Πρέπει να εξετάσουμε όλες τις μεμονωμένες περιπτώσεις και η Κομισιόν πρέπει να καταθέσει μία πρόταση επ' αυτού. Εν τω μεταξύ, μέχρι να γίνει αυτό, εγώ καλώ ε, το ε, Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να έχουν το δικαίωμα έκφρασης βέτο, δικαιώματος αρνησικυρίας. Αν θέλετε, αυτό είναι μια πρόσκληση προς την κατεύθυνση της ε, Κομισιόν. Εγώ καλώ την Κομισιόν αυτές τις ε, προτάσεις ε, προσαρμογής να τις καταθέσει το συντομότερο δυνατόν. όσον αφορά στην έκθεσή μου, έχουν κατατεθεί τροπολογίες από τους συναδέλφους, από συναδέλφους Τσικάου και Αλαγεσέντα η ε, τροπολογία της κυρίας Τσικάο. Εκεί νομίζω ότι υπάρχουν μερικά θέματα που είναι περιτά. Ε, Παραδείγματο χάρη 8 και 9. Εκεί η κυρία Τσικάο ε, αναφέρει ότι θα πρέπει να δημοσιεύονται οι τελικές αποφάσεις των επιτροπών. Μα αυτό έτσι και προβλέπεται στη συνθήκη της Λισαβόνας και ως εκ τούτου κρίνω ότι είναι περιττό. Εξάλλου αυτές οι αποφάσεις δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Δεν είναι λοιπόν απαραίτητο να το επισημαίνουμε εμείς. Όσον αφορά την τροπολογία υπαριθμών 10. Ε, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Επιτροπή Μεταφορών. Ίσως να είναι χρήσιμο για κάποιες άλλες επιτροπές, αλλά δεν αφορά εμάς. Και όσον αφορά την ε, τροπολογία υπαριθμών 12, ε, εκεί η τροπολογία, η κυρία Τσικάο θέλει να γνωρίζει ε, πώς ακριβώς θα παρτίζονται οι επιτροπές. Εγώ λοιπόν προτείνω να μην τοποθετηθούμε από αυτού. Τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που καλούνται να αποφασίσουν ε, για το ποια θα είναι η σύνθεση των επιτροπών. Εξάλλου αυτό είναι σε άμεση συνάρτηση και με το κόστος και μην ξεχνάμε ότι για κάθε επιτροπή μπορούμε να έχουμε τέσσερις εκπροσώπους ε, ανακράτως μέλος. Καλύτερα λοιπόν ας τα αφήσουμε αυτό το θέμα. Η τροπολογία υπαριθμών 13 είναι εντάξει. Αυτή ε, κατά κάποιον τρόπο ταυτίζεται με αυτά που λέω εγώ στην δική μου την υπαριθμών 4. Όσον αφορά την τροπολογία υπαριθμών 18 ε, πρέπει να σας πω ότι εγώ μπορώ να δεχτώ εδώ ε, συμβασμό. Όσον αφορά τι τροπολογίε συναδέλφου 11. υπάρχει η τροπολογία υπαριθμών 11, η οποία σε μεγάλο βαθμό ε, σύμφωνα με τη δική μου την 3, η 17 είναι πολύ καλή. Εκεί η σε θεωρεί και ζητάει το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί τι εξελίξει στα έγγραφα. Μερικέ φορέ λοιπόν ε, έχουμε στην αρχή το σχέδιο του κειμένου και μετά το κείμενο αυτό τροποποιείται σημαντικά. Θα ήταν λοιπόν λογικό να παρακολουθούμε λιγάκι το πώς εξελίσσεται ένα κείμενο. Να μην έχουμε μπροστά μας μόνο το τελικό κείμενο, αλλά και γενικά το πώς προέκυψε το τελικό κείμενο. Αυτά είχα να σας πω εν είδη και παρακαλώ είμαι... Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον ε, συνάδελφο ο οποίος ε, παρουσίασε μια πολύ καλή δουλειά. Εδώ είναι ένα σημαντικό θέμα με το οποίο πρέπει να εξοικειωθούμε αλλά είναι απαραίτητο ε, να εφαρμόσουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας και ως εκ τούτου θα κληθούμε ως βούλευτες να δώσουμε κάποιο νέο ορισμό στις ε, πράξεις κατεξουσιοδότηση και στις εκτελεστικές πράξεις. Αλλά πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε η παλιά διαδικασία της επιτροπολογίας να μην εφαρμόζεται μόνο στις, εκτελεστικές, στις πράξεις κατεξουσιοδότηση και εμεί στις εκτελεστικές πράξεις να μην έχουμε κανένα απολύτως δικαίωμα. Αυτό είναι καθοριστική σημασία. Το πρώτο είναι νομοθετικής φύσεως, έχει σχέση με την Επιτροπή, η Επιτροπή ε, να μπορεί να δραστηριοποιηθεί. Μετά όμως ε, εμείς στις ε, εκτελεστικές πράξεις εκεί πλέον δεν θα έχουμε αρκετές αρμοδιότητες για να ελέγξουμε την Κομισιόν. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο σε αυτή την ειδική επιτροπή που θα υπάρχει, που θα αντικαταστήσει την επιτροπολογία, εκεί τα κράτη-μέλη ε, με τους εμπειρογνώμονές τους θα έχουν δικαίωμα ψήφου και οι Κομισιόν. Εκεί λοιπόν και εμείς να ενημερωνόμαστε παράλληλα χρονικά ε, την ίδια στιγμή με την Κομισιόν, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να ασκήσουμε επιρροή γιατί είναι αλήθεια ότι εμείς ε, ως βουλευτές πρέπει να έχουμε το καθεστώς του παρατηρητή. Μερικές φορές είναι απαραίτητο να υπάρχει φυσική παρουσία, ε, και όχι μόνο να διαβάζει κανείς ε, τα πρακτικά κύριε Πρόεδρε αλλά να γνωρίζει και πώς ακριβώς προέκυψε μία απόφαση. Εμείς λοιπόν ως ΕΛΚ ε, το υπογραμμίζουμε αυτό ακριβώς όπως και τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί και που ο εισηγητής ε, μερικές από αυτές έχει δεχθεί και άλλες πάλι όχι. Υπάρχει περιπτώσει, ο κατάλογος ψηφοφορίας και εκεί μπορείτε να δείτε με τι συμφωνούμε εμείς. Και μία παρατήρηση που αφορά στην μεταβατική περίοδο. Είναι σημαντικό να υπάρχει μία πρόβλεψη, να μην περάσουμε δηλαδή απότομα από την επιτροπολογία σε πράξεις κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές ε, πράξεις. Αλλά και εκεί να έχουμε για κάποια μεταβατική περίοδο τη δυνατότητα ε, διαφωνίας ε, ως ευρωβουλευτές. Μιλάω δηλαδή για δύο μήνες, ένα χρονικό διάστημα που αν κρυθεί απαραίτητο να παραταθεί το διάστημα αυτό με άλλους δύο μήνες. Αυτά είχα να παρατηρήσω και σας ευχαριστώ πολύ για την καλή σας δουλειά ως εισηγητής. κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, νομίζω ο κύριος Αλντράου έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Η επιτροπολογία ε, δεν ήταν πάντα το αγαπημένο θέμα της Επιτροπής Μεταφορών, ούτε και τώρα είναι, έστω και με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι λοιπόν πολύ λεπτή αυτή η δουλειά το να διαπιστώσει κανείς ε, πώς ακριβώς θα εφαρμόζονται θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα του ε, Κοινοβουλίου μέσα από τις ε, πράξεις κατά και τις εκτελεστικές ε, πράξεις. Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση καλούμεθα να γνωμοδοτήσουμε. Η βασική δουλειά θα γίνει στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και εκεί είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν περισσότεροι νομικοί από ό,τι υπάρχουν εδώ. Αυτοί λοιπόν θα προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν το τι περιλαμβάνεται στη συνθήκη της Λισαβόνας ε, και πώς όλα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν για να ενισχυθούν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Νομίζω λοιπόν ότι ορισμένες από τις ε, τροπολογίες κατά την άποψή μας είναι πολύ πιο προχωρημένες από αυτά που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Βεβαίως αυτό είναι θέμα ερμηνείας. Σε πάρα πολλά θέματα ε, συμφωνώ με αυτά που προτείνει ο εισηγητής και όπως ε, σας είπα ανεξάρτητα με το ε, ποιος είναι ο κατάλογος ψηφοφορίας περιμένω να δω τι θα γίνει τελικά με τις διάφορες επιτροπές και κατά πόσο θα υπάρξει ενίσχυση των δικαιωμάτων μας γιατί σε τελική ανάλυση αυτό μας ενδιαφέρει. Σα ευχαριστούμε πολύ. Νόμιζα ότι είχαμε ολοκληρώσει τον κατάλογο των ομιλητών. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ όμως ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το ζήτημα της επιτροπολογίας που έχει το λόγο. Κοιτάξτε, εγώ ε, ασχολούμαι με το θέμα αυτό στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και ως εκ τούτου το ε, παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστώ ευχαριστούμε πολύ για τις ε, τροπολογίες. Είναι ε, ξεκάθαρες, εύκολα εφαρμόζονται ε, και εγώ με μεγάλη μου χαρά θα τις παρουσιάσω και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Εδώ πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, γιατί ως Επιτροπή Μεταφορών δεν πρέπει να υποτιμούμε το θέμα. Πρόσφατα είχαμε την χαρά να ε, εφαρμόσουν τη διαδικασία επιτροπολογίες για τα υγρά που μεταφέρονται στα αεροσκάφη. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η επιτροπολογία και αν δεν προσέξουμε τώρα τότε τα δικαιώματα τα οποία μας αναγνωρίζονται με τη συνθήκη της Λισαβόνας ποτέ δεν θα γίνουν σεβαστά. Γιατί δυστυχώς υπάρχει μια αρνητική τάση τόσο στην Κομισιόν όσο και στο Συμβούλιο να μας περικόψουν τα δικαιώματα αυτά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για πόλεμο και εμείς ως Κοινοβούλιο καλούμεθα να υπεραμεινθούμε του αποτελέσματος ε, της ε, συνθήκης της ε, Λισαβόνας. Γι' αυτό λοιπόν συνάδελφοι μην τα παίρνετε ελαφρά όλα αυτά που αναφέρονται εδώ είναι καθοριστική σημασία για το μέλλον και ειδικά στις τεχνικές προδιαγραφές, στους σαρωτές σώματος, στα υγρά που μεταφέρονται μέσα στα αεροσκάφη. Εκεί λοιπόν κατεβλήθησαν προσπάθειες να να αγνοηθεί ή έστω να υπονομευθεί η άποψη του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν, για αυτά τα δικαιώματα μιλάμε, αυτά τα δικαιώματα που μας αναγνωρίζει η συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Εδώ συμφωνώ με τον συνάδελφο και θεωρώ αυτά που είπατε σχετικά με το καθεστώς του παρατηρητή αυτό είναι καθοριστική σημασία γιατί μόνο με την ε, παρουσία μας θα μπορέσουμε να συμβολήσουμε το ότι ε, υπάρχουν εξελίξεις ε, που μπορούν να επηρεαστούν από το Κοινοβούλιο. Και βεβαίως σε τέτοιου είδους θέματα μπορούμε στην Ολομέλεια της Επιτροπής μας να συζητάμε και να αποφασίζουμε το τι ακριβώς ε, συμβαίνει με αυτές τις ε, πράξεις ε, κατ' εξουεδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις. Σε τελική ανάλυση, σε μας λένε οι ψηφοφόροι μας ότι όλα αποφάσεις παίρνετε και τίποτα δεν γίνεται. Αυτό ακούμε συνέχεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω, Σάιντ, έχεις να προσθέσεις κάτι. Δεν είσαι υποχρεωμένος. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Απλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την υποστήριξη και τα σχόλιά τους. Όντως, είναι κάπως βαρετά αυτά τα θέματα. Κι όμως, τα διαδικαστικά ζητήματα θα είναι πολύ σημαντικά για το έργο μας τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να βάλουμε τα όρια μας. Δεν, μπορούμε να γίνω, δεν επιτρέπεται να γινόμαστε έρμεα των καταστάσεων. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές μας στο έπακρο. Και περιμένω η Νομική Επιτροπή να δείξει πυγμή στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, γιατί είναι δική της αρμοδιότητα και όχι της Επιτροπής Μεταφορών. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο. ή μάλλον πριν να συγχαρώ τους Γερμανούς συναδέλφους για την νίκη τους στο διαγωνισμό της Eurovision. On Saturday. Το Σάββατο. Θα ήθελα να συγχαρώ και τους Βέλγους για την ε, πολύ αξιόλογη παρουσία τους. Και το Ηνωμένο Βασίλειο που πάτωσε δυστυχώς το διαγωνισμό. Βέβαια δεν μπορούμε να αποκλειστούμε τελείω γιατί είμαστε και χορηγοί. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση γνωμοδότηση Βλάσακ για τα πρότυπα και τις επιδόσεις των καινούριων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές. Κύριε Ζήλικ, σας ευχαριστούμε θερμά που είχατε την καλοσύνη να αντικαταστήσετε τον κύριο Βλάσακ στην παρουσίαση της γνωμοδότησης. Υπάρχει διαδικαστικό ίσως για το σύστημα ψηφοφορίας ε, στο διαγωνισμό της Eurovision, κύριε Γκρός. Και εγώ ε, θα ήθελα να συγχαρώ για τη Λένα. Και... Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφασίσουμε σήμερα για την έκθεση αυτή ε, και να συζητήσουμε για τροπολογίες και συμβαστικές προτάσεις. Εμείς πήραμε δεύτερο και τρίτο. Ε, τώρα ήταν και τέταρτο κατάλογο ψηφορίας και είπαν θα έρθει κι άλλος. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω τη συζήτηση για την ψηφοφορία να την αναβάλουμε για την επόμενη συνάντηση και γενικά να πούμε ότι αν κάποιος ε, στην Επιτροπή ε, προσπαθήσει να καταλήξει ε, σε μία συμβαστική πρόταση ε, θα πρέπει να την έχει ανακοινώσει μία μέρα νωρίτερα στους υπόλοιπους για να μπορούν και άλλοι να ασχοληθούν με την πρόταση αυτή. Η γνώμη σας ποια είναι για να μην πάρω μία απόφαση και μετά προκύψουν αντιρρήσεις. Μια στιγμή να διαβουλευτώ. The information I'm getting, Matthew, is that... Matthew. Μου λένε και διορθώστε να κάνω λάθος ότι επισημάνθηκε αυτό στον εισηγητή αλλά δεν θέλει να αναβληθεί περαιτέρω το θέμα. Παρόλο που υπήρχε πρόβλημα με τη διαβίβαση των συμβαστικών τροπολογιών στα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών. Είναι αδιέξοδο κάπως το ζήτημα αν συμφωνεί με την αναβολή ο εισηγητής δεν θα υπήρχε πρόβλημα, αν συμφωνούσε. Αλλά από ό,τι ξέρω δεν βλέπει με καλό μάτι την αναβολή. Βέβαια από εσά εξαρτάται τι θέλετε. Οι σκιώδεις εισηγητές τι γνώμη έχουν μάθει. Äh, Κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, με κάθε σεβασμό προς τους συναδέλφους, αλλά τώρα 5 παρα 5 μου λέτε ότι θα κατατεθούν και άλλες ε, τροπολογίες αργότερα, ε, τότε σήμερα τι να συζητήσουμε αφού δεν έχουμε τελειώσει. Ας δούμε και τη γνώμη των υπόλοιπων εισηγητών. Ο κύριος από το ΕΛΚ, κυρία Βαγιώμα από το ΑΣΔ, Στέρξ, Άλντε, Κράμερ από τους Πρασίνους, και ο Σκιώδης από την ΚΟΕ. Ας κάνουμε ένα μικρό γύρο τραπέζης να βολιδοσκοπήσουμε τους Σκιώδης ηγητέ για το τι προτιμούν. Ντομινίκ. Δεν ξέρω, ο συντονιστής μας ε, τι συμβουλεύει. Α, ασφαλού εσύ. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, Τάνια. Well, Brian, I... Μπράιαν, περιμένω να ακούσω τις προτάσεις των συναδέλφων, αλλά αν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό, τότε θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε, αλλά δεν είναι ξεκάθαρη τοποθέτηση ούτε των σχεδόν εισηγητών και λείπει και ο εισηγητής που είναι πολύ δύσκολο να λάβουμε αυτή τη στιγμή μία απόφαση. Μα και εμένα μου κάνει εντύπωση το ότι δεν είναι εδώ εισηγητής. Είναι πολύ δύσκολο άνευ εισηγητή να γίνει μια συζήτηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση απουσία του. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή εμεί να πούμε αν θα πρέπει να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Πρόεδρος, ναι, αλλά έχει να κάνει αυτό με τις εκλογές στην τσεχική δημοκρατία. Βέβαια αυτό είναι πάντα ένα πρόβλημα γιατί πάντα προκύπτουν κάπου εθνικές εκλογές. Ντέρκ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, αν ε, είναι προβληματική η συζήτηση σήμερα και αν πρέπει να γίνει, ε, αν δεν μπορεί να γίνει ψηφοφορία αύριο. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να εκφράσω την άποψή μου στην πολιτική ομάδα. Ε, πάντως, αν ο Ματιό έχει προβλήματα στην πολιτική του ομάδα, εγώ θα του ασκήσω πίεση. Δηλαδή εγώ θέλω να γίνει και συζήτηση και ψηφοφορία. Μάικλ. Κοιτάξτε, εγώ υποστηρίζω αυτά που λέει ο Μάτιο Εγκρό. Δηλαδή, δεν μπορούμε εδώ να συζητήσουμε για τροπολογίε που δεν γνωρίζουμε. Εγώ τα email ε, δεν τα ξέρω. Ήρθανε 4 παρα 5. Εγώ ήμουν εδώ. Πού να τα δω. Άρα, δηλαδή, να αναβληθεί και η συζήτηση και η ψηφοφορία. Κύριε Γουέλς. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν δύο περίεργα πράγματα. Ένας κατάλογος ψηφοφορίας όπου υποτίθεται ότι θα ψηφίσουμε unblock ε, συνολικά για όλες τις τροπολογίες ενός ανθρώπου και όχι για συγκεκριμένα άνθρωπα. Αυτό είναι πολύ περίεργο γιατί δεν μπορεί κανείς να καταλήξει με τον τρόπο αυτό σε συμβαστικές προτάσεις και εξάλλου ούτε και εγώ είδα συμβαστικές προτάσεις. Κάποιες φήμες άκουσα και νομίζω δεν μπορούμε τώρα να μιλάμε σοβαρά εδώ, να σοβαράμε για φήμες. Τι είναι αυτά. Γι' αυτό και εγώ λέω αναβολή. Ρόμπερτ, θέλεις να πεις τίποτα. Ναι, όσον αφορά το διαδικαστικό τμήμα, δεν γνωρίζω πολύ καλά όλες τι λεπτομέρειες. Ο κύριος ε, Βλάζακ ήδη από το Στρασβούργο μου είχε πει ότι δεν επρόκειτο να έρθει σήμερα λόγω των εκλογών στην Τσεχική Δημοκρατία. Όσον αφορά όμως πληροφόρηση που πήρα από την ομάδα μου, όσον αφορά τον συμβασμό, Νομίζω ότι η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής θα μπορούσε να προχωρήσει σε ένα συμβασμό. Εμείς όμως δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, η δική μου ομάδα τουλάχιστον, και νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν να αναβάλουμε την ψηφοφορία και θα ήταν ιδιαίτερα ευγενικό οξυνόματος των άλλων πολιτικών ομάδων να μας επιτρέψουν να βολεί αυτή. Πρόεδρος, από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρος πρέπει να αποφασίσει τελικά. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, σαφή, πολύ ωραία. Λοιπόν, άκουσα τις απόψεις όλων. Είναι σαφές ότι το ζήτημα είναι σημαντικό και όντως υπάρχουν κάποιες πολιτικές ομάδες που λένε ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν πλήρως συμβαστικέ προτάσεις και δεν είναι σε θέση να ψηφίσουν λοιπόν αύριο. Και δεν βοηθά βέβαια καθόλου το ότι απουσιάζει και ο εισηγητής. Καταλαβαίνετε όμως πώς έχει κατάσταση, όταν έχουμε εθνικές εκλογές συμβαίνουν αυτά. Συνεπώς, σα προτείνω να αναβάλουμε την συζήτηση και την ψηφοφορία για την έκθεση αυτή μέχρι την επόμενη συνάντησή μας και μέχρι τότε θα καταφέρουμε να βρούμε λίγο χρόνο στα πλαίσια του χρονοδιάγραμματός μας για να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Συγγνώμη, Ρόμπερτ, εσείς θέλετε να προχωρήσετε, έπρεπε εγώ όμως να πάρω μια απόφαση και δεν θα μπορούσα να πάρω μια απόφαση όπου υπάρχει μια σημαντική πολιτική ομάδα που λέει όχι, άλλε ομάδε λένε όχι, οι σοσιαλιστέ λένε όχι ή ίσω. Προτείνω λοιπόν, δεδομένων όλων αυτών, να αναβάλουμε τη συζήτηση και την ψηφοφορία μέχρι την επόμενη, τον επόμενο μήνα, side. Μια γενική παρατήρηση. Αυτό που είπε ο Μάθιου είναι σωστό. Είναι πολύ δύσκολο να εργαστεί κανείς όταν λαμβάνει τελευταία στιγμή τις συμβαστικές προτάσεις. Πριν από μια ψηφοφορία πρέπει κανείς συζητήσει και με συναδέλφους από άλλες πολιτικές ομάδες. Επομένω, θα ήταν καλό να είχαμε κάποιε κατευθυντήρε γραμμέ και για του συζητητέ όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Ξέρω δεν υπάρχουν γενικοί κανόνε επ' αυτού και μερικέ φορέ καλείται κανεί στο τέλο μια διαδικασία να κινηθεί πολύ γρήγορα, αλλά ωστόσο σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να... Μάλλον δεν θα μπορεί να γίνει ποτέ ψηφοφορία απουσία του εισηγητή. Εκτό και αν συμφωνούμε όλοι για όλα, αλλά όταν η κατάσταση είναι συγκεχημένη όπω και σήμερα, τότε είναι απαραίτητη η παρουσία, σου, η παρουσία του. Πρόεδρο, ακριβώ επειδή το ζήτημα είναι τεχνικό, ακριβώ επειδή χρειαζόμαστε τον εισηγητή, ακριβώ επειδή έχουμε τόσε πολλέ τροπολογίε, χρειαζόμαστε την εμπειρογνωμοσύνη του εισηγητή. Γι' αυτό το λόγο σκέφτηκα και εγώ ότι είναι καλύτερα να περιμένουμε μέχρι τον ερχόμενο μήνα. Και δεν νομίζω ότι θα ήταν και πολύ ε, δίκαιο για τον εισηγητή να προχωρήσουμε απουσία του γιατί θα έπρεπε να είναι σε θέση να απαντήσει σε ενδεχόμενες παρατηρήσεις ή ερωτήσεις των συναδέλφων. Γι' αυτό το λόγο σας προτείνω να αναβάλουμε την όλη διαδικασία μέχρι τον επόμενο μήνα και ζητώ από τη Γραμματεία τον επόμενο μήνα καταφέρει να βρει τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να γίνει συζήτηση και η ψηφοφορία της έκθεσης αυτής. Θα προχωρήσουμε έτσι κατεξαίρεση αυτή τη φορά λόγω των συνθήκων των της Ας πάμε στο επόμενο σημείο τώρα. Πιο γρήγορα φτάνουμε σε αυτό από ό,τι περιμέναμε. Θα μιλήσουμε για τους σιδηρόδρομους και για την εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους και για την αξιολόγηση, εκτίμηση τροπολογιών, τροποποίησεων όσον αφορά αυτή την πρώτη δέσμη. Αυτό είναι το θέμα μας να ευχαριστήσω καταρχάς τους συντονιστές που μου ζήτησαν να καταλήξω σε ένα ψήφισμα μετά την προφορική ερώτηση. Και βλέπω μετά ότι οι πολιτικές ομάδες υπέβαλαν πάρα πολλές τροπολογίες βέβαια σε αυτό το οποίο πρότεινα. Το σχέδιο ψηφίσματος που έχετε Προσπάθησα να το κάνω όσο πιο ισορροπημένο γίνεται, δηλαδή να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στα ζητήματα που περιγράφονται εδώ για τους σιδηροδρόμους και το ζήτημα τη μη συμμόρφωση των κρατών μελών και τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το ζήτημα. Καταλαβαίνω ότι ορισμένε από τι τροπολογίε που υποβλήθησαν έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο χρειαζόμαστε για του σιδηροδρόμους. και συμφωνώ ότι όντω πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και να επέλθουν πολλές βελτιώσεις στο σιδηροδρομικό σύστημα. Το ψήφισμα όμως αυτό έχει να κάνει πιο συγκεκριμένα με την εφαρμογή μιας συγκεκριμένη νομοθεσίας. Θα ήθελα να πω λοιπόν στους αδέλφους από την Ανατολική Ευρώπη ότι εγώ θα είμαι παρόν σε οποιαδήποτε διαδήλωση γίνει, σε οποιαδήποτε κινητοποίηση γίνει προκειμένου να καταφέρατε να εξασφαλίσετε περισσότερη χρηματοδότηση για τους σιδηροδρόμους σας. Θα είμαι πάντα μαζί σας αυτά τα αιτήματα. Επαναλαμβάνω όμως ότι αντικείμενο της έκθεσης αυτής δεν είναι η υποδομή των σιδηροδρόμων, δεν είναι η περαιτέρω χρηματοδότηση για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Η συγκεκριμένη εντολή που μου δόθηκε είναι να αξιολογήσω την εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους και πιο συγκεκριμένα να αναφερθώ στο ζήτημα της μη συμμόρφωσης των κρατών μελών. Σας το λέω λοιπόν αυτό από την αρχή για να τα πράγματα ξεκάθαρα. Τώρα, το ψήφισμά μου επικεντρώνεται στο ότι δεν γίναν σπουδαία πράγματα τα πέντε τελευταία χρόνια για την εφαρμογή της πρώτης αυτής δέσμης απουσία επίσης ε, ανάληψης δράσης όχι μόνο από τα κράτη-μέλη αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρομαι επίσης στο ότι δεν ήταν ανεξάρτητοι πάντα οι ε, διαχειριστές των σιδεροδρομικών υποδομών. Επίσης ότι δεν υπήρξε ο απαραίτητος έλεγχος για τις συνθήκες ανταγωνισμού και ότι δεν ικανοποιητικό το σύστημα των τελών για τους σιδηροδρόμους. Στο τέλος της πρότασης ψηφίσματος λέγεται ότι θα πρέπει να αναθωρηθεί η πρώτη δέσμη μέτρων το 2010, ότι αυτό αποτελεί σημαντικότατη προτεραιότητα και λέγεται επίσης στο ψήφισμα ότι θα πρέπει να επιληθούν τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα και ότι θέλουμε την πλήρη εφαρμογή και συμμόρφωση με το πακέτο αυτό και ότι αυτό αποτελεί εκ των ουκ άνευ προκειμένου να λειτουργήσει σωστά το συνδρομικό δίκτυο στην Ευρώπη. Έχουν υποβληθεί 47 τροπολογίες που έχουν να κάνουν κυρίως με την χρηματοδότηση των σιδεροδρομικών υποδομών. Ορισμένες άλλες τροπολογίες που συμπεριλήφθησαν έχουν αποδυναμώσει το ψήφισμα γιατί διαγράφουν τις αναφορές που γίνονται στα κράτη-μέλη που δεν συμμορφώνονται ή διαγράφουν τις ε, επικρίσεις που γίνονται όσον αφορά το ότι δεν λειτουργούν οι απαραίτητοι κανόνες ανταγωνισμού, ορισμένοι ζητούν την απόλυτη απελευθέρωση του στεροδρομικού δικτύου και για τη μεταφορά των επιβατών αν όχι αμέσω τουλάχιστον στο εγγύ μέλλον. Υπάρχουν άλλε τροπολογίε που έχουν να κάνουν με την ανεξαρτησία των διαχειριστών υποδομών και ορισμένοι συνάδελφοι ζητούν περισσότερε πληροφορίε για τι νομικέ ερμηνείε που υιοθετεί από τη μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την άλλη τα κράτη-μέλη. Και υπάρχουν και πάρα πολλέ τροπολογίε που έχουν να κάνουν με, τις, με τα τέλη για τι υποδομέ. Ορισμένοι επικρίνουν το, τα, τους χαμηλούς διαθέσιμους πόρους και υπάρχουν άλλοι που επικρίνουν την ε, μη εφαρμογή και τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς, της πρώτης δέσμης δηλαδή μέτρων. Βλέπουμε επίσης ότι έχουμε πλέον 22 χώρες με την συμπερίληψη της ε, Βουλγαρίας που έχουν ε, εφαρμόσει την πρώτη δέσμη μέτρων που έχουν αρχίσει να την υλοποιούν. Αρχικά θα θυμάσαι ότι είχαμε 21 μόνο χώρε. Ω πρόεδρο τώρα τη επιτροπή μας και έχοντα λάβει εντολή από εσά, θα ήθελα καταρχάς να έχουμε μια γενικότερη συνένεση σε επίπεδο ε, επιτροπής, με συγχωρείτε, όσον αφορά το ψήφισμα και ξέρω ότι υπάρχουν ζητήματα που δεν θα είναι αρεστά σε μια πολιτική ομάδα και άλλα ζητήματα με τα οποία δεν θα, συμφωνεί, άλλη πολιτική ομάδα. Αυτό το οποίο θέλω να πετύχω είναι να πετύχουμε μια γενικότερη ευνοϊκή θέση για το ψήφισμα και θα πρέπει να λέμε συνολικά ότι το θεμελιώδες ζήτημα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι ότι 22 κράτη-μέλη δεν έχουν εφαρμόσει την πρώτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους και ότι αν είναι να προχωρήσουμε περισσότερη απελευθέρωση των σιδηροδρόμων και αν θέλουμε τελικά να έχουμε ένα αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα, τότε αν μη τι άλλο θα πρέπει να, αρχίζουμε, να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε την πρώτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Και γι' αυτό το λόγο είπα ότι ε, σαφώς θα μπορούσαμε όλοι να συμπεριλάβουμε επιμέρους τεχνικά ζητήματα τα οποία θα θέλαμε να βελτιωθούν στους εθνικούς σιδηροδρόμους, αλλά είναι καλύτερο να τα ξεχάσουμε όλα αυτά τα τεχνικά ζητήματα και να πούμε καταρχάς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς τα κράτη-μέλη ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι η πρώτη δέσμη δεν έχει εφαρμοστεί και ότι δεν έχει αναλυφθεί νωρίτερα δράση για να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. και να αναφερθώ και σε αυτό το οποίο υπόθηκε το ότι όντως οι, σιδηρόδρομοι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις προκειμένου να βελτιωθούν και προκειμένου να εφαρμοστεί τελικά η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Θα το συμπεριλάβω και αυτό στο ψήφισμα, ότι αν όντω θέλουμε να βελτιώσουμε τους σιδηροδρόμους, τότε όντω θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις από τα κράτη-μέλη προκειμένου να βελτιωθούν οι σιδηρόδρομοι και να εφαρμοστεί η πρώτη δέσμη. Δεν θα ήθελα όμως και πάλι να καταλήξουμε σε μία κατάσταση όπου θα δίνονται γενικά δικαιολογίες για ποιο λόγο τα κράτη-μέλη δεν εφάρμοσαν την ε, πρώτη δέσμη μέτρων. Γιατί πριν από μερικά χρόνια και τα κρατημέλη συμφώνησαν μαζί μα για αυτή την πρώτη δέσμη. Επομένω, α μην του δίνουμε τώρα δικαιολογίε για ποιο λόγο δεν εφάρμοσαν αυτή την πρώτη δέσμη. Σα ευχαριστώ για τι τροπολογίες σα, Προσπάθησα να κρατήσω μια ισορροπία στα πλαίσια του ψηφίσματο και θα ήθελα στο τέλος της διαδικασίας, όταν επισήμωση υποβάλλουμε το ψήφισμα, να είναι, σαφές πλέον, να είναι σαφής πλέον η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε να εφαρμοστεί, να υλοποιηθεί η πρώτη δέσμη μέτρων και θέλουμε να ληφθεί απαραίτητη δράση προκειμένου να αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα με τα οποία συμφωνήσαμε πριν από μερικά χρόνια. Κύριε Γκρός, έχετε το λόγο. Ε, Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε συστήσει επανειλημμένα για το θέμα αυτό και έχει φτάσει πια η χρονική στιγμή να εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε αποφασίσει εδώ και χρόνια. Και νομίζω εκ μέρους του ΕΛΚ μπορούμε να πούμε ότι ε, σε πολλά θέματα θα συμφωνήσουμε. Στα σημαντικότερα μάλιστα. Και νομίζω όσον αφορά με μονομένες ε, τροπολογίες θα ε, συμφωνήσουμε μαζί σας. Ο κύριος Μαρνέσκου ε, το είπε πολύ διπλωματικά, είπε να μην αναφέρεται ο, αναφέρονται ονομαστικά τα κράτη. Εμείς λέμε όχι να αναφέρονται καλύτερα. Εξάλλου υπάρχουν χώρες όπου υπάρχει διαχωρισμός ε, ανάμεσα ή διαχωρισμός και διαφοροποίηση όσον αφορά την υποδομή των ε, σιδηροδρόμων. Και αυτό μάλιστα με υποστήριξη της Κομισιόν. Θεωρούμε όμως στο ΕΛΚ ότι αυτό δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να καταλήξουμε στην επιλογή κάποιων όρων που θα έδινε ε, το επιχείρημα σε άλλα κράτη-μέλη να προβούν σε τέτοια ερμηνεία ώστε να πούνε «Α, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ανεξαρτησία των διαχειριστών υποδομής». Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα υποστηρίξουμε τη δική σας την πρόταση και γνωρίζοντας ότι για μας ο διαχειριστής ε, ε, της υποδομής ε, θα πρέπει να είναι παντελώς ανεξάρτητος γιατί κατά παρελθόν διαπιστώσαμε ότι αν Οποτεδήποτε δεν υπήρξε διαχωρισμός ρυθμιστικών φορέων και διαχειριστών υποδομής, δημιουργήθηκαν προβλήματα. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε ε, πρώτα απ' όλα τι θα γίνει με το πρώτο πακέτο πριν φτάσουμε στο δεύτερο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να ε, προβούμε σε κάποιες, να δεχθούμε κάποιες παραλήψεις και μετά να πούμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Εμείς είμαστε υπέρ του ανοίγματος της αγοράς, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. το υπογραμμίζω αυτό. Ο καταναλωτής είναι εκείνος ε, που θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό μας μέλημα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται πραγματικά να προσφέρονται με σωστό τρόπο. Αυτό βέβαια δεν είναι κατά του ανοίγματο της αγοράς. Εγώ του αντίον θεωρώ ότι μια ένα λογικό ανοίγμα της αγοράς μπορεί να ωφελήσει τον καταναλωτή και ε, οικονομικά στέκεται επίσης. Εξάλλου, αυτό που δεν μπορούμε να δεχθούμε είναι ότι ορισμένα κράτη να αρνούνται το άνοιγμα της αγοράς. Από την άλλη όμως οι επιχειρήσεις τους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς ε, στο ε, εξωτερικό. Ε, αυτό δεν θέλω τώρα να πω λεπτομέρειες. Καλή είναι αυτή στο Παρίσι, αλλά τώρα, το Δεκέμβρη του 2009, το ΕΡΑΤΕΠΕ να κατοχυρώνει ε, το μονοπόλιο του χωρίς καμία αντίδραση, συγγνώμη, Ντομινίκ, και απ' την άλλη να λέει ότι στη Ρώμη μπορεί κανείς να συμμετέχει στον δημόσιο διαγωνισμό. Γι' αυτό λοιπόν, Πρόεδρε, παρακαλώ, στον ε, συμβιβασμό, στον οποίο καταλήξαμε μετά από συζήτηση στην πολιτική μας ομάδα. Παρακαλώ λοιπόν αυτή την συμβαστική πρόταση να την υποστηρίξουμε, εκεί να προβλέπετε η αρχή της αμοιβαιότητας. Γιατί δεν είναι δυνατόν εμείς να βοηθάμε τους άλλους, εκείνοι να μην ανοίγουν την αγορά τους και αυτοί να μπορούν να συμμετέχουν στους δημόσιους διαγωνισμούς τρίτων, όπου το επιτρέπει αυτό η ε, νομοθεσία. Αυτή είναι η θέση της, ε, του ΕΛΚ. Νομίζω είναι και πιο αμβλημένη σε σχέση με το παρελθόν ε, και σε γενικές γραμμές εμείς διατηρούμε τη θέση μας. Γι' αυτό λοιπόν όπως σας είπα, θα υποστηρίξουμε την πρόταση του εισηγητή. Ευχαριστώ, Μάθιο. Ο κύριος Αλκαντράου για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, μετά ο κύριος Στέρξ. Θα μας δώσουν τη βελγική προοπτική του θέματος. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ μαζί σας ότι στο ψήφισμα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου. Γιατί μπορούμε να μιλούμε εκτενώς για τους σιδηροδρόμους. Θα μπορούσαμε μέχρι και πολυσέλιδο έργο να συγγράψουμε. Αλλά θα πρέπει να επιμείνουμε στο άνοιγμα των αγορών και στην εφαρμογή του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου. Και με το ψήφισμά μας να διαβιβάσουμε ένα κατηγορηματικό μήνυμα. Φυσικά δεν θα πρέπει να μακρηγορήσουμε σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία των διαχειριστών των υποδομών. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία τους. Θα απορρίψουμε οποιαδήποτε τροπολογία που προσπαθεί να σχετικοποιήσει ή να περιορίσει αυτή την ανεξαρτησία. Εγώ θα υποβάλω τροπολογίες για τη χρηματοδότηση. που συνδέονται με το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο. Το σύστημα, για παράδειγμα, εισφορών για να δημιουργηθούν κονδύλια που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα για τη χρηματοδότηση, για να εξασφαλιστεί το μέλλον των σιδηροδρομικών μεταφορών, που μας ενδιαφέρει όλους. Σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, θα γνωρίζετε ότι ούτε η πολιτική μου ομάδα εκθιάζει την απελευθέρωση. Υπάρχουν βέβαια πλεονεκτήματα στο άνοιγμα των αγορών, αλλά δεν είναι για μας η ιερή αρχή. Θα πρέπει να συνοδεύεται η απελευθέρωση με αποτελεσματική διαλειτουργικότητα, με την εξασφάλιση των κοινοφελών υπηρεσιών και μια λύση για τη χρηματοδότηση των σιδηροδρόμων. Δεν θα δώσουμε το πράσινο φως σε κάτι που θα περιορίζεται μόνο στο εμπορικό στοιχείο της απελευθέρωσης, την οποία θα χαρακτηρίζει ως πανάκια. Εμείς είμαστε υπέρ του ανοίγματο των αγορών και για τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Αρκεί να εξασφαλιστεί μεγαλύτερο μερίδιο των μεταφορών εμπορευμάτων από τους σιδηροδρόμους. Αυτό για μας είναι σημαντικό, να αυξηθεί το μερίδιο των σιδηροδρόμων στη μεταφορά εμπορευμάτων. Αλλά τώρα μιλάμε περισσότερο για τις μεταφορές επιβατών. Τι θα γίνει λοιπόν από εδώ και πέρα. Για να συνεχίσουμε στο άνοιγμα των αγορών θα πρέπει να εφαρμόσουμε το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο. Συμφωνώ με τον κύριο Γκρό για την αμοιβαιότητα. Έχει απόλυτο δίκιο. Και οι χώρες που έχουν επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα σε τρίτες χώρες θα πρέπει εφαρμόζοντας συνεργείς αμοιβαιότητες και οι τρίτες χώρες να ανοίξουν τις αγορές τους. Δεν μπορεί κάποιος να προστατεύει την αγορά του και να εποφθαλμιά παρόλα αυτά την αγορά και του γείτονά του. Αυτά ευχαριστώ. Κατά του λοιπόν συμφωνώ με τον πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριο Στέρξ από τους φιλελεύθερους. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Και εγώ και εγώ συμφωνώ με την πρότασή σας ότι χρειαζόμαστε ένα κείμενο για την εφαρμογή του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου. Γιατί δεν μιλούμε ούτε για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ούτε για τη χρηματοδότηση των κοινοφελών υπηρεσιών. Για αυτά τα θέματα θα ακολουθήσουν άλλα ψηφίσματα. Εδώ μιλούμε για την εφαρμογή του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου. Έχει παρέλθει μία δεκαετία από την έγκριση αυτού του πακέτου και διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών εξακολουθεί να μην το εφαρμόζει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γίνει μια συζήτηση για αυτό το πακέτο. Ένα πακέτο που εγκρίθηκε πριν από 10 χρόνια, αλλά συνεχίζουμε τη συζήτηση για την ερμηνεία του. Άλλο επικροτεί την αλφα ερμηνεία και άλλο προτιμά τη διτερμηνία. ερμηνεία. Θα πρέπει να πιέσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε το συντομότερο δυνατό να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτό το πακέτο. Δίκιο έχει ο ΣΑΙΤ. Φυσικά είναι σημαντική η διαλειτουργικότητα. Αν όμως το μόνο που καταφέρουμε είναι να διωγγώσουμε την γραφειοκρατία, να διαχωρίσουμε τις υπηρεσίες, να δημιουργήσουμε μια ρυθμιστική αρχή. Όλα αυτά είναι προϋποθέσεις που δεν έχουν νόημα αν δεν συνοδεύονται από άνοιγμα των αγορών. Και στόχος αυτού του πακέτου είναι το άνοιγμα των αγορών, ώστε ένας πάροχος μιας χώρας να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε άλλη χώρα. Και μάλιστα να γίνεται αυτό με εύρυθμο τρόπο. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον αποτελεσματικά ή ισορροπημένα. Κάποιες χώρες έχουν καταφέρει να κρατήσουν στο περιθώριο αυτή τη στιγμή τους αντιπάλους τους και ή de facto ή de jure να διασφαλίσουν το κρατικό μονοπόλιο. Οι σιδηροδρομικές ε, αγορές δεν είναι υγιείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό συμφωνώ με την πρόταση του Προέδρου. Να δεχτούμε το πακέτο και να το εφαρμόσουμε το συντομότερο δυνατό, χωρίς περικοκλάδες. Και να επιμείνουμε στο άνοιγμα των αγορών, με τον α β τρόπο. Και ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι στείλαμε mail και απάντηση δεν λάβαμε. Τι γίνεται με την τροπολογία 46. Στην τροπολογία 46 λέμε ότι αν δεν υλοποιηθεί το άνοιγμα των αγορών, όλα αυτά τα μέτρα θα αυξήσουν τη δημοκρατία, την γραφειοκρατία και θα είναι περιτά. Τι γίνεται με την τροπολογία μου 46 για το άνοιγμα των αγορών, δεν έλαβα απάντηση για τη τύχη της. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ νομίζω ότι είσαι λίγο αυστηρός, Μπράιν. Ε, Εντάξει, το καταλαβαίνω, ως δάσκαλος πρέπει κανείς να είναι αυστηρός. Αλλά το γεγονός ότι περιορίζεται τώρα μόνο σε αυτό το πρώτο πακέτο σιδηροδρόμων. Κοίταξε να δει. Ε, εδώ ασκούμε κριτική στην Κομισιόν. Η νομοθεσία έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και 10 χρόνια και η Κομισιόν περίμενε να δει τι θα κάνει. Παρότι βέβαια γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παραλήψει εδώ και χρόνια. Και ε, βεβαίως, ε, εδώ η κριτική που ασκούμε προς την Κομισιόν συνοδεύεται και από τότε έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό. Δεν μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε τα μάτια τι ακριβώς συμβαίνει σε άλλους τομείς, γιατί η Κομισιόν μεταξύ άλλων έχει το καθήκον να επιβάλλει τον δίκαιο ανταγωνισμό στους σιδηροδρόμους. Αν συνεχίσει αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός, ο τομέας των σιδηροδρόμων μπορεί να είναι τέλειος, μπορεί να υπάρχει πολύ, καλή, πολύ καλός διαχωρισμός ε, των ε, παρόχων και των δικτύων, αλλά η Κομισιόν δεν θα έχει καμία ευκαιρία να παρέμβει, γιατί, ε, παραδείγματος χάρη, θα είναι φτηνή οι σιδηρόδρομοι, αλλά θα είναι ακριβά τα διόδια ή αντίστροφα. Γι' αυτό λοιπόν δεν καταλαβαίνω το ότι την δική μας την τροπολογία, την υπαριθμόν 28, την απορρίπτεις. Μα αυτή η τροπολογία απλά επισημαίνει ότι η Κομισιόν πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα. Ούτε εγώ τώρα θέλω να ξεκινήσω ολόκληρη συζήτηση για τον αθέμητο ανταγωνισμό, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε, ε, γιατί αυτό ισχύει για την Κομισιόν εδώ και χρόνια. Τώρα, ο ανταγωνισμό, όπως είπαμε, παίζει καθοριστικό ρόλο και γι' αυτό πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκε πλαίσιο. Η διαφορετική πρακτική που ανέφερε ο συνάδελφο αναφέρεται και αυτό σημαίνει ότι ε, όλες αυτές οι χώρε που αναφέρονται δεν μπαίνουν όλες στο ίδιο καζάνι. Υπάρχουν μεγάλε διαφορέ ανάμεσα στη Γερμανία και τη Γαλλία. Το και εσύ. Ε, στην Γερμανία εγώ τότε παρουσίασα το πρώτο πακέτο σιδηροδρόμων και εκεί αναφέρεται ότι οι χώρες οι οποίες έχουν προετοιμαστεί εδώ και χρόνια για να ανοίξουν τα δίκτυά τους αυτές οι χώρες επέφεραν σημαντικά αποτελέσματα 60% ε, στην Ολλανδία ή στην Πολωνία 25% αύξηση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών στη Γερμανία όλες αυτές οι χώρες λοιπόν που ήταν κλειστές αυτές τελικά βίωσαν μία μία μείωση της τάξης του 28% που σημαίνει ένα 28% ε, των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών μεταφέρθηκε στους δρόμους και αυτό πρέπει να το πει κανείς και στα συνδικάτα της Γαλλίας ε, που κατεβαίνουν στους δρόμους τι κάνουν, μποϊκοτάρουν τα ξένα βαγόνια για να μην χάσουν ε, τη δουλειά τους. Αυτή είναι μια αλήθεια που πρέπει να την πούμε. Και η αμοιβαιότητα βεβαίως είναι ένα καθοριστική σημασία κριτήριο το οποίο εμείς πάντα το αναφέραμε. Και εάν λοιπόν υπάρχει οποιοδήποτε εμπόδιο τότε ε, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ξεχάσουμε το θέμα του δίκαιου ανταγωνισμού. Κοιτάξτε γιατί. Εάν μία εταιρεία λαμβάνει απευθείας ανάθεση με μια τιμή που δεν μπορεί όμως να συγκριθεί, τότε θεωρητικά αυτή η επιχείρηση μπορεί να λάβει μια παραγγελία, ένα έργο με αύξηση της τιμής κατά 30%. Και με αυτό το 30% μπορεί κανείς όταν είναι στο εξωτερικό να κατέβει γιατί θα το πάρει το 30% πάλι στην πατρίδα του. Αυτή η έλλειψη αμοιβαιότητας καταστρέφει τον ανταγωνισμό. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς είμαστε υπέρ του διαχωρισμού του δικτύου και του παρόχου. Ξέρουμε ότι αν αυτά υπάρχουν στον ίδιο ε, φορέα αυτό οδηγεί στην κατάχρηση. Απαραίτητη η αμοιβαιότητα. Ως εκ τούτου λοιπόν πρέπει να υπάρχει κάποιο συμβασμό, Brian, να αναφέρεται οπωσδήποτε η αμοιβαιότητα. Αλλιώ μπορούμε να το ξεχάσουμε το όλο θέμα. Α δούμε λοιπόν γιατί είμαστε υπέρ του ανταγωνισμού και υπέρ του ανοίγματο των δικτύων. Να σα αναφέρω ένα παράδειγμα από τη Γερμανία. Εκεί οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι πριν από 10 χρόνια είχαν το μονοπόλιο και ήθελαν να κάνουν τη διαδρομή να πάυσουν μια διαδρομή κάπου εκεί στο Ντούσελντοφ με την αιτιολογία ότι χρησιμοποιείται αυτή η γραμμή μόνο από 500 επιβάτες την ημέρα. Όμως ε, οι ενδιαφερόμενοι τα χωριά δεν το ήθελαν αυτό, ε, προκήρυξαν διαγωνισμό και ο νέος επενδυτής ε, σκέφτηκε, κανονικά έπρεπε να συμμετέχουν οι σιδηρόδρομοι και τι είχε διαπιστώσει αυτός ο άνθρωπος, ότι δεν υπήρχε διαλειτουργικότητα. Μόλις έφτανε το τρένο είχε φύγει το λεωφορείο. Αυτός λοιπόν, ο νέος επενδυτή, άλλαξε λιγάκι τα ωράρια και μέσα σε 10 χρόνια διαπιστώθηκε μία αύξηση από 500 σε 20.000 επιβάτες την ημέρα. Αν δεν υπήρχε ο ανταγωνισμός και αν ε, τα πράγματα τα ρύθμιζε μόνο του το μονοπόλιο, είτε είναι κρατικό είτε όχι, θα είχε πάυσει να υπάρχει εκεί συνδρομική διασύνδεση και αυτοί οι 20.000 άνθρωποι θα κυκλοφορούσαν με τα αυτοκίνητά τους. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να το αποφύγουμε και το κίνητρο πρέπει να είναι πάντα ότι ε, δεν αποφασίζει μόνος του κανείς αν θα κλείσει μια γραμμή όχι. Μπορεί να, το, να αναλάβει κάποιος άλλος, ο οποίος μάλιστα μπορεί και να επωφεληθεί από αυτό. Να πω και κάτι άλλο. Αναφέρομαι στη δική μας την τροπολογία, την υπαριθμών 28, την οποία δυστυχώς θέλει να απορρίψει ο εισηγητής. Επ' αυτού λοιπόν να πω το εξή όσον αφορά τις συνθήκες πλαίσιο. Κοιτάξτε, όσον αφορά την 28 καταρχήν. Στην Ευρώπη έχουμε 30 δις ευρώ που ε, λαμβάνουν, ε, που είναι στις τσέπες των αεροπορικών εταιριών γιατί δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Αυτό λοιπόν για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στη πρέπει κάπως ε, να μπορούν να το εξοικονομήσουν η Σλοβακία τι έκανε. Επέβαλε διόδια στους σιδηρόδρομους, στις εμπορευματικές μεταφορές. Διπλάσια από τη Γερμανία. Και κατάργησε τις, ε, τα διόδια στους δρόμους καλή αυτή η κίνηση αλλά προς λάθος κατεύθυνση. Γιατί λοιπόν είμαι εγώ υπέρ της τροπολογίας παριθμών 26, γιατί αν εγκριθεί 25 του κύριου Κούνε, καταπίπτει 26. Πολλά πράγματα είναι ίδια σε αυτές τις δύο, αλλά ένα πράγμα διαφέρει. Εμείς στη δική μας την τροπολογία ζητάμε να υπάρχουν ε, διαφανή συστήματα τιμολόγησης. Γιατί επιμένω σε αυτά. Γιατί στη Γερμανία έχουμε μια κατάσταση όπου στο Βερολίνο έχουμε ένα τιμολόγιο για τις αστικές μεταφορές που είναι διπλάσιο από ότι σε άλλες περιοχές. Μέχρι τώρα λοιπόν κανείς δεν μπόρεσε να μου εξηγήσει γιατί να ισχύει κάτι τέτοιο. Και για αυτό το λόγο χρειαζόμαστε να υπάρχει διαφάνεια στις τιμές. Δεν είναι δυνατόν στο Βερολίνο ε, οι σιδηρόδρομοι να πίνουν το αίμα του κράτους, να αποφασίζουν μόνοι τους να αυξάνουν τις τιμές και σε άλλα μέρη πάνε αλλού ε, και κάνουν ε, φτηνότερες προσφορές. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι η τροπολογία η υπαριθμών 26 παρακαλώ να παραμείνει ακόμα και αν εγκριθεί η τροπολογία υπαριθμών 25 την οποία και στηρίζουμε. Δεν είναι όμως όλα ίδια, αυτό ήθελα να πω. Και εγώ επιμένω η ε, τροπολογία 26 να παραμείνει και η 28 είναι σαφές ότι εμεί εστιάζουμε την προσοχή μας στο πρώτο πακέτο των σιδηροδρόμων. Αλλά α μην ξεχνάμε ότι κοιτάμε και πέρα από τη μύτη μας. Ε, τώρα, μια τροπολογία μπορεί να γίνει δεκτή χωρίς εδώ να χρειαστεί ε, να ξεκινήσουμε ατέρμονες συζητήσεις για τη διλατουργικότητα. Νομίζω ότι γίνεται αυτό ε, και παρακαλώ πολύ να δεχτείτε την τροπολογία υπαριθμών 28. Um, uh, um, Ο κύριος Ζήλ. Γενικώ το κόμμα μας ε, οι μεταρρυθμιστές και συντηρητικοί είναι υπέρ της δικής σας προσέγγισης, υπέρ του πλήρους ανοίγματος των αγορών με εφαρμογή του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου. Βέβαια, όπως θα είδατε, μόνο μία τροπολογία καταθέσαμε, την 39, δικής μου έμπνευσης, και θα ήθελα να επισύσω την προσοχή σας στην τροπολογία αυτή που δίνει ένα πολιτικό μήνυμα γιατί έχουμε και γεωγραφικά, ιστορικά και εμπορικά ζητήματα που δεν είναι παρόμοια σε όλα τα κράτη-μέλη. Και στο θέμα των βαλτικών χωρών, εκεί οι μόνες εταιρείες προς τις οποίες μπορεί να, ανοίξει, να ανοίξουν οι αγορές είναι ρωσικές. Οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι. Πριν από λίγε ε, εβδομάδες είχαμε τον κύριο Γιακούνιν εδώ για πρόγευμα εργασία στις Βρυξέλλες και εξέφρασε ενδιαφέρον να έρθει στις αγορές των βαλτικών χωρών. Αλλά θα πρέπει να καταλάβει τα χαρακτηριστικά των σιδηροδρομικών μεταφορών στις Βαλτικέ χώρες. Αν υπήρχε θεσμικός διαχωρισμός των εταιριών στις σιδηροδρομικέ μεταφορές θα γίνουμε πολύ ευάλωτοι και τρωτοί στο μέλλον. Ιδιαίτερα με αλλάξει η πολιτική κατάσταση και η κατάσταση αγοράς. Πριν από δύο-τρία χρόνια είχαμε παρόμοια κατάσταση στην Εστονία με την, με την καταδάφιση ενός μνημείου σταμάτησαν οι εμπορικές μεταφορές από τη Ρωσία ως αντίπινο. Το ίδιο είχαμε και με την περίπτωση ενός ε, αγωγού πετρελαίου. Όταν δεν έλαβαν οι Ρώσοι αυτά που ήθελαν από εμά, ε, μπλόκαραν την διέλευση πετρελαίου. Την περασμένη φορά αναφέρατε το παράδειγμα της Φιλανδίας. Εγώ πάντως από τις εμπειρίες μου που έχουμε τους λετωνικούς σιδηροδρόμους, διαπίσω ότι η Φιλανδία και η Εστονία έλαβαν πολλές εξαιρέσεις από το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο. Δεν είμαι βέβαια η Δήμον στα θέματα αυτά, δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες. Ίσως από νομική άποψη η Φιλανδία έχει πολύ μεγάλες διαφορές από ότι οι βαλτικές χώρες για την εφαρμογή του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου. Πάντως θα ήθελα να λάβετε υπόψη ότι η αγορά στις βαλτικές χώρες είναι πολύ διαφορετική. Δεν μιλάμε για αγορές Βελγίου, Γερμανίας ή άλλων χωρών που είναι παρόμοιες. Οι δικές μας αγορές είναι πολύ διαφορετικές στις βαλτικές χώρες. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη και το πολιτικό υπόβαθρο κάποιων αποφάσεων που θα λάβει σε τέτοιο εμπορικό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριο Σκούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι μας ε, ποια κατεύθυνση θέλουμε να ακολουθήσουμε. Θέλουμε στην Ευρώπη να έχουμε κοινή αγορά σιδηροδρόμων. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν ε, στοιχεία στην κοινή αγορά όπως η αμοιβαιότητα. Να υπάρχει λοιπόν ε, αμοιβαιότητα, αυτό είναι καθοριστική σημασία, ε, να συμμετέχουν όλοι κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όταν θα έχουμε επιτύχει να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός των φορέων, τότε είναι απαραίτητο εκείνοι που συμμετέχουν στον ανταγωνισμό ε, σε αυτούς να μπορεί κανείς να αναλύσει τις δομές και πώς ακριβώς επιδοτούνται αυτοί οι φορείς. Αυτό είναι καθοριστική σημασία για να μην προκύπτει στρέβλωση του ανταγωνισμού, να μην ε, υπάρχουν ε, συγκαλυμμένες επιδοτήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη έτσι ώστε οι τιμές των εισιτηρίων να είναι σαφείς, διαφανείς και από την άλλη πλευρά να υπάρχουν και ξεκάθαροι όροι σχετικά με τις προκηρύξεις διαγωνισμών. Κύριε Στέρξ, έχετε να σχολιάσετε κάτι ακόμη. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση για τον κύριο Αρχαντραουή. Στην τροπολογία 31 που συνδυάζεται με την τροπολογία 28 του κυρίου Κράμερ, αν και υπάρχουν μικρές διαφορές μεταξύ των δύο. Στην Ολλανδική μετάφραση, το πρωτότυπο είναι στα αγγλικά, αλλά στην ε, Ολλανδική μετάφραση δεν βγάζω νόημα από την πρώτη φράση. Θα πρέπει να υπάρξει σύγκληση των αρχών ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες θεμητού ανταγωνισμού. Τι εννοείται ακριβώς. Μήπως ουσιαστικά κάνετε αυτό που λέει και ο κύριος Κράμερ στη δική του τροπολογία. Γιατί ο κύριος Κράμερ λέει ότι μπορούμε να επιβάλλουμε τέλη, ιδιώδια, παρόμοια με των οδικών μεταφορών, για να υπάρξει ίση μεταχείριση σιδηροδρομικών και οδικών. Αν όντω είναι αυτή η πρόθεσή σας, θα στοιχήσει πολύ στους σιδηροδρομικού φορείς. Βέβαια το πρωτότυπο είναι αγγλικά, κύριε Καντραουή. Ευχαριστώ. Αυτό που εννοώ είναι ότι θα πρέπει να θεσπίσουμε κριτήρια που θα ισχύουν για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Τώρα για το πώς θα εφαρμοστούν θα πρέπει να το εξετάσουμε. Θέλουμε να υπολογιστεί εσωτερικά το εξωτερικό κόστος όλων των τρόπων μεταφοράς. Δηλαδή σε κάποιο βαθμό να υπάρξει σύγκληση. Σύγκληση προς ένα ενιαίο σύστημα χρέωσης. Αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και άλλες πτυχές. Στην αεροπορία, για παράδειγμα, στις αερομεταφορές, καταβάλλεται ΦΠΑ. Στους σιδηροδρόμους επιβάλλεται τέλος ηλεκτρισμού, για παράδειγμα. Διαφέρουν όμως οι επιβαρύνσεις ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς. Ίσως προτρέχουμε, ίσως ε, παρά είναι διεξοδικό αυτό το επίπεδο και λεπτομεριακό. Ας ε, χαράξουμε κάποιες ε, γενικές γραμμές για το μέλλον. Ναι, ναι. Και βλέπω ότι συμφωνεί και ο εισηγητής, ο πρόεδρος, ο κύριος Κράμερ. Ο εισηγητής συμφωνεί επί της ουσίας, αλλά όχι με τον τύπο. Ή όλοι θα πληρώνουν το φόρο πετρελαίου, είτε κανένας. Ή κανένας δεν πληρώνει. Αυτή τη στιγμή οι σιδηρόδρομοι καταβάλουν φόρο ρηκτό καυσίμων. Οι οδικές μεταφορές το ίδιο. Η αεροπορία όχι. Αν πάω με τρένο από το Βερολίνο στις Βρυξέλλες, δεν είναι ότι θα χάσω τρει φορές περισσότερο χρόνο, είναι ότι θα πληρώσω και τριπλάσιο εισιτήριο. Γιατί είναι πολύ υψηλότερα τα τέλη στι μεταφορέ από ό,τι στι αερομεταφορέ. Άλλο ισχύει στις ναυτιλιακές μεταφορές. Τα σιδηροδρομικά εισιτήρια είναι πολύ πιο ακριβά. Επιβάλλονται τέλη που είναι υποχρεωτικά. Αν εξετάσουμε το θέμα της εμπορίας εκπομπών, για παράδειγμα. Τα θέματα του ηλεκτρισμού στους, στους σιδηροδρόμους. Είναι πολύ ψηλό το τέλος ηλεκτρισμού που καταβάλλονται από τους σιδηροδρόμους. Κάτι που αποβαίνει βάρος του σε σχέση με την αεροπορία που τη χάνει ευνοϊκότερης μεταχείριση. Εγώ αυτό που ζητώ είναι ίση μεταχείριση για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Γιατί να πληρώνουν τα σπασμένα μόνο οι σιδηρόδρομοι. Στη Γερμανία κάθε όχημα επιχορηγείται, επιχορηγείται περίπου 3.000 ευρώ το χρόνο. Αν όλα υπολογιστούν εσωτερικά, τότε θα είναι πολύ πιο ακριβώς ο σιδηρόδρομος και αυτές τις διαφορές της θέλουμε να καταργήσουμε. Ναι, αλλά επιχορηγήσεις υπάρχουν παντού. Γι' αυτό είναι τόσο φτηνά μερικές φορές κάποια εισιτήρια. Μάλλον έκανα λάθος, λέει ο πρόεδρος. Ίσως εγώ διέπραξα λάθος, γιατί προσπάθησα να βολέψω όλες τις ομάδες και τελικά βρήκα τον πελά μου. Γιατί όλοι θέλουν να είναι πιο φιλόδοξοι τώρα ξαφνικά. Έπρεπε εγώ να ήμουν πιο αυστηρός από την αρχή και να περιοριστώ στο πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο τελεία και παύλα. Εγώ φταίω που προσπάθησα να ακούσω τις εκκλήσεις των συντονιστών και να καταρτήσουμε ένα ψήφισμα μετά τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Εν πάση περιπτώσει και σερά σερά, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει στην ψηφοφορία, αλλά για τη συγκεκριμένη ερώτηση ως προς την τροπολογία 46. Άλλαξα γνώμη, γιατί νομίζω ότι η τροπολογία 46 καλύπτεται από τη συμβαστική λύση Α Μπορεί να διαφωνείτε, αλλά εγώ πιστεύω ότι η συμβαστική πρόταση Α, α τη βρω μέσα σε αυτό το χαρτομάνι, λέει κάτι παρόμοιο με τη δική σας τροπολογία 46. Θεωρεί ότι το επιτυχημένο άνοιγμα των αγορών στις σιδηροδρομεταφορές θα εξαρτηθεί από την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου περαιτέρω απελευθέρωση τη αγορά σιδηροδρόμων θα πρέπει να αποβεί βάρο τη ποιότητα των σιδηρομεταφορών και θα πρέπει να διασφαλίζονται οι κοινοφελεί υπηρεσίε στου σιδηροδρόμου. Μπορεί βέβαια να μην είναι τόσο κατηγορηματική διατύπωση με τη δική σα, αλλά επί τη ουσία νομίζω ότι καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία. Ρόμπερτ, μίλησε για τη Λιθουανία. Όντω, η Ανατολική Ευρώπη έχει ιδιαίτερα προβλήματα επιπλέον. Τώρα για τη Φιλανδία. Δεν νομίζω ότι χέρι εξαίρεση ιδιαίτερη ή ειδικών προνομίων. Θα το ερευνήσω πάντως. Δεν θέλω όμως να έχουμε ένα πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο με 22 εξαιρέσει. Ε, αυτό θα είναι σιδηροδρομικό πακέτο μόνο για 5 χώρε άμα 22 τη χάνουν για να μην πω καν πέντε, γιατί η Μάλτα και η Κύπρος δεν έχουν σιδηροδρόμους. Αυτό φοβάμαι με την δική σου πρόταση. Καταλαβαίνω το πρόβλημα και μάλιστα πήγα στη Φιλανδία ακριβώ για να εξετάσω το ζήτημα μας, ιδιαίτερα για τα θέματα των διασυνοριακών ζητημάτων με την Ρωσία. Και οι σιδηρόδρομοι για τις βαλτικές χώρες είναι πολύ σημαντική. Τώρα, αν έχουμε μια ειδική λύση για Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία, και άλλες χώρε χώρες θα ζητήσουν για μεταχείριση για άλλα επιμέρους ζητήματα. Και τα τελευταία 20 χρόνια αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Πάντα βρίσκουν προσχήματα οι σιδηρόδρομοι για να δημιουργήσουν κολλήματα και να παρεμποδίσουν την πρόοδο. Όλο αυτό συμβαίνει. Και εγώ πραγματικά αγαπώ του σιδηροδρόμου και μακάρι να σημειωθεί πρόοδο. Δεν μιλάω μόνο για αυτό που είπατε εσεί, αλλά πολλοί προσπαθούν να, βάλουν εμπόδια στο, στο δρόμο τη πρόοδου για του σιδηροδρόμου τα τελευταία χρόνια. Όπω είπα, και σερά σερά. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Και αυτό τραγούδι από την Eurovision δεν ήταν ή επηρεάστηκα από το Σάββατο. Η Doris Day το είχε πει. Ποιο το είχε τραγουδίσει, τέλο πάντων. Θα αποφασίσει η Επιτροπή μας, θα δούμε τι θα αποφασίσει και μετά θα προχωρήσουμε. Ό,τι και να αποφασίσει η Επιτροπή πάντως, ο ρόλος μας Πρόεδρο είναι να τον υπερασπίσω στην Ολομέλεια, ακόμη κι αν καταρρύπτεται η προσωπική μου γνώμη. Μέρος του καθήκοντος του Προέδρου είναι να προσπίσει τη θέση της Επιτροπής, άσχετα με τις προσωπικές του απόψεις. Πάντως, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι είχαμε πάρα πολύ καιρό, είχαμε, ήμασταν πολύ μπροστά στο πρόγραμμα μέχρι που φτάσαμε στους σιδηροδρόμους. Εκεί που είχαμε κερδίσει ένα σωρό ε, ώρα με τη διεκπαιρέωση των, των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, με το που μπήκαμε στους σιδηροδρόμους κολλήσαμε. Εκεί όλοι θέλησαν να μιλήσουν, ναι θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο, αλλά ένα σωρό προβλήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εκεί που ήμασταν μπροστά στο χρόνο μας, τώρα βρεθήκαμε να μένουμε και πίσω. Άλλοι λένε νέα απελευθέρωση, αλλά απελευθέρωση τώρα. Άλλοι λένε απελευθέρωση νέα, αλλά αργότερα. Αυτά τα προβλήματα έχουμε. Πάντα όταν μιλούμε για τους σιδηροδρόμους, όλοι είναι κατενθουσιασμένοι, λατρεύουν τους σιδηροδρόμους, αλλά με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Και φάνηκε αυτό και στις συζητήσεις που είχαμε και χαίρομαι που είναι συναρπαστική συζήτηση και εξάπτονται τα πάθη, γιατί πραγματικά η σιδηρόδρο, είναι θεμελιώδης κλάδος και χαίρομαι που υπήρξε τέτοια σφόδρη συζήτηση. Μία ακόμη ερώτηση για την τροπολογία 26. Δεν καταπίπτει με την έγκριση της 25. Λάθος το αναφέρει ο κατάλογος ψηφοφορίας. Καλώς θα το ελέγξουμε, Μάικλ, ποια θα είναι η τύχη της τροπολογίας 26 αν η 25 εγκριθεί. Θα το εξετάσει η γραμματεία. Πάντως το βλέπω με καλό μάτι. Θα το, θα το εξετάσουμε. Ωραία. Εντάξει. Διακοπή της τακτικής συνεδρίασης. Θα συνεδριάσουν οι συντονιστές τώρα. Θέλετε αμέσως ή διάλειμμα. Ρόμπερτ, είσαι έτοιμος. Ωραία. Okay.